I, Is there anybody who lost this yesterday evening? Δεν ξέρω αν ε, κάποιος ε, ξέχασε κανείς κάτι εδώ. Καλαμάτζη. Ναι, ήταν εδώ ίσως, είναι Ιταλικό. Ποιανού είναι αυτό. Μάλλον δικό του είναι, καλώς. Εν πάση περιπτώσει, εάν δεν ε, βρίσκεται σήμερα εδώ, θα το κρατήσει η γραμματεία για τον κύριο Καλαμάτζη, γιατί νομίζω σε αυτόν ανήκει. Καλημέρα λοιπόν. Ελπίζω η πρώτη μέρα της συνεδρίασής μας να μην αποδείχθηκε πολύ δύσκολη για σας. Ε, συνεχίζουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξή μας. Περνάμε στο σημείο 6 ε, αυτής όπου έχουμε να προβούμε σε ψηφοφορία σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Έχουμε τροπολογίες οι οποίες είχαν υποβληθεί από τη δική μας από την Επιτροπή ε, και άρα αυτή τη στιγμή μπορούμε να συζητήσουμε ε, τις τροπολογίες της δικές μας, της δικής μας Επιτροπής και η συνάδελφος Helga Trippel είχε να λάβει να υποστηρίξει τις δικές μας τροπολογίες, τα δικά μας συμφέροντα. 59 ε, συνολικά τροπολογίες από τους συναδέλφους μας κατατέθηκαν και όσες από αυτές τώρα τις τροπολογίες ε, περάσουν θα υποβληθούν στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Η Επιτροπή Προϋπολογισμών θα αξιολογήσει τις τροπολογίες αυτές και εφόσον τις εγκρίνει και εκείνη θα ε, υποβληθούν πλέον στην Ολομέλεια. Θα ήθελε η Helga Trüppel να πει κάτι έτσι προκαταρκτικά. Ευχαριστώ, Ντόρις. Ε, για τα νέα λοιπόν εδώ μέλη της Επιτροπής ε, θα ήθελα να πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά το πώς έχουν τα πράγματα και το γιατί εγώ είμαι εισηγήτρια, ήμουν και είμαι εισηγήτρια. Λοιπόν, από την τελευταία βουλευτική θητεία, η οποία ήταν και η πρώτη για μένα στο Κοινοβούλιο, ε, είμαι, ήμουν μέλος εδώ της Επιτροπής και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών από την πλευρά των Πρασίνων και ήμουν και συντονίστρια για τη δική μου πολιτική ομάδα και πάντα εγώ είχα υποστηρίξει ε, την αναβάθμιση της ε, ευρωπαϊκής ε, πολιτικής πολιτισμού και της ευρωπαϊκής πολιτικής παιδείας γιατί, αλλά και γενικά το μέσο, γιατί βέβαια αν δεν έχουμε για παράδειγμα και κινηματογράφο, ο οποίο είναι ευρωπαϊκό και σε διάφορε γλώσσε, τότε δεν μπορούμε να δώσουμε και το κατάλληλο ένωσμα, τα κατάλληλα κίνητρα για την ευρωπαϊκή διάσταση. Οπότε το είναι το υπόβαθρο από το οποίο εγώ δραστηριοποιούμε εδώ, αλλά βέβαια και δραστηριοποιούμε και στην Επιτροπή των Προπολογισμών, αλλά εδώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ε, όπως θα είδατε, ε, κατατέθηκαν ένα σωρό διαφορετικές ε, τροπολογίες, γιατί έτσι έχουν εδώ τα πράγματα, μόλις μας εξήγησε και η Doris Πακ. Δηλαδή, η Επιτροπή αρχές του έτους ή τέλος πάντων μέχρι το καλοκαίρι προβαίνει στη σύνταξη του πρώτου σχεδίου του προπολογισμού, το Συμβούλιο εξετάζει αυτό το σχέδιο και ε, πολύ συχνά προβαίνει σε διαγραφή ε, συγκεκριμένων ε, γραμμών του προπολογισμού, πράγμα βέβαια που μα εκνευρίζει επανειλημμένα γιατί ειδικότερα σε τομείς όπως τα μίντια, όπως ο πολιτισμός, όπως η παιδεία είναι πάρα πολύ σημαντικά αν θέλουμε να προσεγγίσουμε και τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο της πολιτικής επικοινωνίας και γι' αυτό αυτό που εμείς προτείναμε είναι ουσιαστικά να επανέλθουμε στην αρχική πρόταση, στο αρχικό δηλαδή προσχέδιο προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά συνέπεια κατάργηση των διαγραφών που πρότεινε το Συμβούλιο. Αυτό συνήθω είναι το παιχνίδι ε, που παίζεται εδώ μεταξύ των ε, θεσμικών οργάνων. Δηλαδή έρχεται το Συμβούλιο και λέει ότι επιθυμούμε να δαπανίσουμε λιγότερα κονδύλια και μετά επανέρχεται το Κοινοβούλιο και λέει όχι, είναι σημαντική αυτή η τομή, χρειαζόμαστε τα λόγω κονδύλια. Αυτό είναι το, ε, το σκεπτικό. Σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες λοιπόν ε, οι οποίες ε, προτείνουν ακριβώς να επανέλθουμε στην πρώτερη ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο σχέδιο δηλαδή προϋπολογισμού της, ε, θα τις ψηφίσουμε unblock, όπως λέμε δηλαδή από κοινού όλες μαζί, γιατί δεν έχει νόημα να τις συζητούμε ξεχωριστά. Το συζητήσαμε και με τους συντονιστές ότι όλες οι πολιτικές ομάδες συμφωνούν ούτως ή άλλως. Και από εκεί και μετά έχουμε μία σειρά από ε, τροπολογίες με τις οποίες φτάσαμε σε μια συμφωνία με τους ε, συντονιστέ και τους κοιόδης εισηγητέ. και θα ε, δείτε τώρα, θα εξετάσουμε αυτήν την, αυτόν τον κατάλογο και θα ψηφίσουμε μία προ μία τις εν λόγω τροπολογίες. Πρόεδρος, Ωραία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν σε δύο τμήματα. Θα γίνει σε δύο τμήματα τη ψηφοφορία. Στι πρώτε τέσσερι σελίδε εδώ, το καταλόγου ψηφοφορία, 30 τροπολογίε τις οποίε θα ψηφίσουμε συλλογικά. Το λέω εκ των προτέρων για να το... για να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Κυρία Κούτσον, για το λόγο. Μάρλε, και desearía retirar las enmiendas 58-37. Θα ήθελα να ε, αποσύρω τις τροπολογίες που έχω βάλει 58-37, ε, 58-58 και 58-60. Okay? Okay. Okay. Okay. It's yours. Ah, yes. Please take it. Thank you. Δικό σας είναι, κύριε Καλαμάτζη. Ε, please, nehmen Sie voting list. Ωραία λοιπόν, έχετε μπροστά σας εδώ τη λίστα, Οι πρώτες λοιπόν τέσσερις σελίδες ουσιαστικά αφορούν σε αξίωση των κονδυλίων που είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κατά συνέπεια κατάργηση το προτινόμενη διαγραφή αυτό το κονδυλίων από το Συμβούλιο. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν, υπέρ αυτών των τροπολογιών. Ποιοι είναι κατά. Κανείς, αποχές, ούτε αποχή λοιπόν, άρα συμφωνούμε εδώ ομόφωνα. Τώρα, περνάμε στις επιμέρους τροπολογίες, δηλαδή οι οποίες θα εξεταστούν μία προς μία. Περνάμε στην τροπολογία 5822. Ψήφι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Κανεί. Αποχές. Κανείς. 58-65. Μίλαν Μον. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχέ. Μία αποχή. 58-66 Μπελέτ Πακ Τελάνγκε. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Oral amendment. Από τον συνάδελφο Μπέλετ. Ε, κύριε Μπέλετ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπάρχει μια μικρή αλλαγή στην ε, παρατήρηση, είναι απλώς ε, μια φράση που είναι η υποστηρίζει την δημιουργία προγραμμάτων ε, τοπικών σε διασυναριακές περιοχές και διαμέσου των συνόρων. Για να έχουμε και τις άλλες ομάδες. Ευχαριστώ. Καταλάβατε όλοι. Έχετε, είσαστε εναντίον, υπάρχει κάποιος που να έχει αντίρρηση, όχι. Ιδαλλιώς ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε για την προφορική τροπολογία του κυρίου Μπένετ. Ποιος είναι υπέρ, ποιος είναι κατά. Πέντε κατά και οι υπόλοιποι υπέρ. 5, 8, 5, 6, 5, 8, 6, 7, Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Προφορική τροπολογία. Παπα-Νικολάου. Σκούρια. Ποιος θέλει να εξηγήσει την τροπολογία. Ναι. Σκούρια. Παπα-Νικολάου. Is not here. Δεν είναι εδώ ο Παπα-Νικολάου. Δεν έχουμε χρόνο, δεν έχουμε χρόνο να περιμένουμε, ναι κύριε Σκούρια. Πείτε μας τι έχετε να πείτε. Ε, τροπολογία κυρία Πρόεδρε. And ε, I read the text, the final text.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 paragraph 4 and 6 could be combined with the following version. The contact points could agree a number of measures to fight theft. Τα σημεία επαφής θα συμφωνήσουν για όλα μέτρα. Ένα από αυτά τα σημεία επαφής με κοινή συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών θα είναι το σημείο επαφής με μερικούς γείτονες. Ich habe eine Frage, Herr, Herr Skurier und Herr, Herr Κύριε Σκουλέτη, κύριε Γιώργο, κύριε ένα ερώτημα. Τι εννοείται με, με κλοπή, ενεργό κλοπή, υποτιθέμενη κλοπή πριν από πολλά χρόνια. Τι εννοείται, τι εννοείται με κλοπή, με το theft. Πραγματική κλοπή ή κάτι το οποίο ίσως ίσως έλαβε χώρα 100 χρόνια πριν. Can you explain... Μπορείτε να μας εξηγήσετε με το τι εννοείτε με το κλοπή. Βεβαίως κυρία Πρόεδρε. Η αρχαιοκαπηλεία και στις μέρες μας αποτελεί ένα διεθνές φαινόμενο το οποίο χρήζει άμεση αντιμετώπιση. Είναι μια κατεξοχήν διεθνής εγκληματική πρακτική και μόνο ως τέτοια πρέπει να την αντιμετωπίζουμε. Η ειδική αναφορά σε εκτός ευρωπαϊκής χώρες Μεσογείου γίνεται γιατί τα κράτη αυτά αφενός είναι συχνά στόχος των αρχιακοαπείλων και αφετέρου αποτελούν δίωδο διακίνησης κλεμμένων αρχαιοτήτων. Και εχθές τροποποιήσαμε την τροπολογία μας ώστε να εξαλειφθούν κάποια ζητήματα επικάλυψης συναρμοδιότητας ειδικά με την Ιντερπολ. Και γι' αυτό έχετε σήμερα μπροστά σας τη διορθωμένη εκδοχή. Και ε, επί της ουσίας η τροπολογία στοχεύει στην ενίσχυση των κοινών δράσεων για τον περιορισμό φαινομένων κλοπής τα οποία ε, φαινόμενα παρατηρούμε συνεχώς την τρέχουσα περίοδο. Δεν είναι ένα παλαιό φαινόμενο, είναι κάτι που βρίσκεται σε εξέλιξη. Um Οπότε σα αντιλαμβάνομαι σωστά όταν λέω ότι έχουμε να κάνουμε ενεργό κλοπή. Δεν έχουμε να κάνουμε το παρελθόν. Ωραία, για να είμαστε προσεκτικοί. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ε, παλιό εδώ ε, αρχαίο ή οτιδήποτε άλλο. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας καταλάβαμε. Αντιληπτό για όλους λοιπόν. Ποιο είναι λοιπόν υπέρ αυτή τη τροπολογία, παρακαλώ με ανάταση χειρό. Ποιοι είναι υπέρ. So. Yeah, we have, we have 13. 13. Once again. Ξανά, ξανά να μετρήσουμε. Only 12 PPE. 12 PPE, who is against? 12 άλλοι λοιπόν. Ποιοι είναι τώρα κατά. 12 προς 12. Άρα απορρίπτεται. Τι είπατε? Απορρίπτεται, απορρίπτεται. 12 προς 12 ψήφους, απορρίπτεται. Σε ποια περνάμε τώρα?

11 against and 12 in favor. It's adopted. 11 κατά 12 υπέρ, άρα εγκρίνεται. Μπέλετ Πακ και Σμιτ 58-58 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58-48 Φίζα Αξέλα. Α, καταπίπτει αυτή. Πάντα η Κουτσέτη και αυτή καταπίπτει και αυτή του συγητή επίση, τη συγκητρια μιλαμε Μιλάμε μόνο 58-55 ψήφοι υπέρ. Ψήφι κατά. Δεκατρεις λοιπόν έναντι 7 άρα υπέρ Μιλάν μόνο εξέλαφή σα. Κύριε Μιλαμόν, θέλετε να μας εξηγήσετε λίγο. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μία μικρή προφορική, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Δηλαδή, το κείμενο παραμένει το ίδιο, απλώς δεν αναφέρεται στο συγκεκριμένο, δεν αναφέρεται το συγκεκριμένο κύριο όνομα που αναφερόταν στην αρχική τροπολογία. Δηλαδή, δηλαδή δεν αναφερόμαστε στην κομποστέλα, το υπόλοιπο κείμενο παραμένει για να μην υπάρξουν συγχύσεις και να υπάρξει ευρεία συνένεση. Ε, είμαι επιφυλακτική θα πρέπει να πω και αν διαγραφεί αυτή η αναφορά παρόλα αυτά ε, παραμένει η πρόθεση. Δηλαδή να μην, ε, να μην έχουμε την ίδια σαφήνεια στο κείμενο. Άρα λοιπόν ε, η δική μου επιφύλαξη παραμένει. Κατά συνέπεια δεν μπορώ να συμφωνήσω στη συγγήτρια. Ποιοι είναι υπέρ μάλλον ρώτησε. Πρόεδρος ήταν δυστυχώς εκτός μικροφώνου. Against. Ψήφι κατά. 13 against 4. 5. 13 4, 5, 6. Άρα 13 ενάντια 6. Αγκρίνεται. 58-45 Μανέσκου. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Πλειοψηφία ήταν υπέρ. Λοιπόν. 58-46 Άρα εγκρίνεται πράγματι. Πρέπει να ψηφίσουμε και την επόμενη 58-24 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 58-39 58-39 Κουτσέτ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Εγκρίνεται. 58-25 της εισηγήτριας. Έχετε ζητήσει το λόγο, παρακαλώ. Ε, ε, μήπως μπορείτε να ρωτάτε για αποχές, ε, γιατί... Γιατί πάντα εδώ και 10 χρόνια που είμαστε σε αυτή την επιτροπή μας ζητάνε έτσι, για τις αποχές. Να καταγράφονται και αποχές, γιατί θα ήθελα να απόσχω. 58-25 λέει η πρόεδρος, ψήφι υπέρ ψηφικάτα κατά. Αποχές. Κανείς. 58-43. Εντάξει, είπαμε μια αποχή. 58-43 Λόκεγκάρτ. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Κανείς. Αποχή κύριος Μάρτιν. Εγκρίνεται. 58-17 της συγκήτριας ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58-42. Όχι, καταπίπτει 58-20 της εισηγήτριας. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη καταπίπτει. Και η μεθεπόμενη. Άρα πάμε στη 58-41. Λόκεγκαρτ. Ψήφι υπέρ ψήφι κατά αποχές εγκρίνεται 58-27 της συγκήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58-18 ψήφι υπέρ 58-28 διορθώνεται η Πρόεδρος 58-28 ψήφι υπέρ κατά α, αποχές εγκρίνεται 58-18 καλός, κατά, αποχές, Αγκρίνεται. Προφορετή τροπολογία, Μιλάν Μόν. Απλώς, στα σχόλια αναφέρεται ο Καναδάς και μιλάμε για αύξηση κονδυλίων για μελέτες της ΕΠΑ και τον Καναδά. Ε, πιστεύω δηλαδή ότι θα πρέπει να δούμε αυτό το θέμα της συμπερίληψης του Καναδά. Υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές. 5823. Ψήφι υπέρ. Ψήφι κατά. Αποχές 5862. Υπέρ. Κατά. φτωχές εγκρίνεται. 58-37. Μαρία. Α, είπατε ότι αποσύρατε, μάλιστα, τις 58-37 58-60, ωραία. Πολύ ωραία. Περνάμε τώρα στην ε, προφορική τροπολογία του κ. Μπέλετ. Όχι. Α, α, ωραία. Τι ωραία. Τελειώσαμε. Και αυτή είναι πρώτα όλα είναι, όλα τα έχουμε τακτοποιήσει, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη μας ψηφοφορία, ίσως λίγο άγνωστη διαδικασία για κάποιους από εσά, αλλά την επόμενη φορά νομίζω θα είναι πιο δύσκολη, λέει ο Πρόεδρος. Ας μιλήσω τώρα και πάλι γερμανικά, λέει ο Πρόεδρος. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης σας διάταξης. Στο 7 λοιπόν. Σημείο 7 της σημερινής σας διάταξης. γνωμοδότηση από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής που θα ε, τροφοδοτήσει την ε, σχετική έκθεση της Επιτροπής των Τροπολογιών. Έχουμε λοιπόν εδώ το σχέδιο γνωμοδότησης. Η συντάκτρια του σχεδίου, η κυρία Χέλγα Τρούπολ, μπορεί να μας την παρουσιάσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτήν την σύντομη έκθεση, ε, αυτό που κάνουμε είναι ουσιαστικά να αναφέρουμε εκ νέου τις δικές μας πολιτικές προτεραιότητες στην Επιτροπή των Προϋπολογισμών. Όχι δηλαδή μόνο αναφέρουμε μία σειρά από ψηφία, από κονδύλια τα οποία επιθυμούμε, αλλά αναφέρουμε και τις πολιτικές προτεραιότητες των όσων θέλουμε να επιτύχουμε. Το πρώτο ε, ζητούμενο είναι αυτό που αναφέρθηκε μόλις τώρα ότι δηλαδή ε, αντιτιθέμεθα στις ε, περικοπές που προτείνει το Συμβούλιο και ε, καταβάλουμε τα επιχειρήματά μας γιατί θεωρούμε πως κάτι τέτοιο είναι απαράδεκτο. Δηλαδή οι περικοπές αυτές που προτείνονται από το Συμβούλιο όπως προτείνονται στους όλους αυτούς τους τομείς που αναφέραμε δηλαδή στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στην παιδεία, στην κοινωνία των πολιτών και ούτω καθεξής. Επίσης, στο τμήμα 3β του προϋπολογισμού που ήδη χρηματοδοτείται με πολύ λίγα κονδύλια έχουν και πάλι γίνει ε, περικοπές ειδικότερα σε ό,τι αφορά ε, τα κονδύλια για τους πολίτες και την προβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο ευρύ κοινό. Και κάτι τέτοιο για μας είναι απαράδεκτο ειδικά αν σκεφτεί κανείς και τα χαμηλά, πολύ χαμηλά ποσοστά συμμετοχής και στις εκλογές, προσέλευση στις κάλπες δηλαδή στις ευρωπαϊκές εκλογές. δεν μπορούμε να ενθαρρύνουμε έτσι τους πολίτες μας περικόπτοντας τα κονδύλια τρίτο τώρα ε, σημείο που θα ήθελα να θίξω, κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει μέσα στα επόμενα χρόνια, αλλά και για τη συζήτηση που θα κάνουμε σε λίγο με την κυρία Βάλστρομ, είναι πώς επικοινωνεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς επικοινωνούν τα τρία μεγάλα θεσμικά όργανα, δηλαδή ε, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη δική μου άποψη, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα εδώ. Θα πρέπει να είναι σαφής η corporate identity μας και θα πρέπει να την περάσουμε με πιο ευκρινή τρόπο ε, στους πολίτες μας, δηλαδή ε, κατά πόσο είναι απαραίτητος ο συντονισμός μεταξύ εθνικής και υπερεθνικής δημοκρατίας για να τον αντιλαμβάνονται οι δικοί μας πολίτες, γιατί δεν είμαστε εμείς Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και πρέπει να το διευκρινίζουμε αυτούς τους πολίτες μας, ώστε να κινητοποιούνται και να συμμετέχουν σε όλο αυτό το ευρωπαϊκό project, στο ευρωπαϊκό έργο. Ε, και βέβαια θέλουμε να τους ε, κοινοποιήσουμε και τα όσα κάνουμε για, αυτούς, για αυτούς και όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην πολιτική επικοινωνία. Θέλουμε λοιπόν γι' αυτό ακριβώ το λόγο να ενημερωνόμαστε και τακτικά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τα όσα κάνει για την επικοινωνία με του πολίτε. Εκεί λοιπόν στο σημείο 4 έχουμε σε αυτό το πρόγραμμα πριν ακριβώς ε, ένα κομμάτι των κονδυλίων τα οποία προορίζονται για την πολιτική επικοινωνία ε, και εκεί ε, ε, βλέπουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε και με τις επιμέρους αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διάφορες χώρες ώστε να μπορέσουμε να εμπλέξουμε περισσότερο τους πολίτες στις εκάστορες χώρες. Στο σημείο 5 τώρα έχουμε να κάνουμε με την επικοινωνία την, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους τομείς όπως της εκπαίδευσης, ειδικότερα με τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα από τον κύριο Μιλάν Μον, δηλαδή να αφαιρθούμε για μία ακόμα φορά στην ε, υπερατλαντική μας συνεργασία και από εκεί και μετά αναφερόμαστε ότι το πολιετές ε, πρόγραμμα θα ξεκινήσει το 2011 και γι' αυτό στην πολιτική, την audiovisual, ήχου και εικόνας και στο κινηματογράφο θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δεν ε, μπορούμε να αναφερόμαστε μόνο σε βιβλία ως προς το που προς τα που καθιστόμαστε ως Ευρώπη, ποιες είναι οι διαμάχες μας, ποια είναι τα προβλήματά μας, αλλά από εκεί και μετά χρειαζόμαστε πέρα δηλαδή και από βιβλία και ε, κινηματογράφο και συνεργασία με τρίτες ε, χώρες και έχουν ξεκινήσει ήδη πολύ επιτυχημένα προγράμματα και σε συνεργασίε με άλλε χώρε όπω είπαμε και θέλουμε να συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται όλα στο σημείο 6. Άλλωστε είδαμε πω τα όσα έκανε σε αυτό το πεδίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα τελευταία χρόνια ήταν όλα πολύ θετικά και θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η δουλειά. Ευχαριστώ, Ντόρι. Η πρόεδρο είχε το λόγο, αλλά δεν ακούσαμε. Συμμερίζομαι τα όσα ελέγχθησαν από την κυρία Τρούπελ Μόνο στην παράγραφο 3 θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την σύνταξη. Εκφράζει την ανησυχία του έναντι της ε, υψηλής αποχής κατά τις τελευταίες εκλογές. Νομίζω ότι σε κάθε διεξαγωγή εκλογών όσον αφορά τις ευρωεκλογές υπάρχει ολοένα και υψηλότερη αποχή. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να ερμηνεύσουμε και νομίζω ότι θα πρέπει να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την μία αύξηση της συνολικής συμμετοχής στις τελευταίες εκλογές. Γιατί από το 79 μέχρι σήμερα έχουμε χάσει ένα 20% συμμετοχής. Νομίζω λοιπόν ότι η σύνταξη είναι λιγάκι ατυχής εδώ. Βασικά αυτό μας λέτε ότι θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ειλικρινείς. Ε. Εντάξει, ε, καταθέστε εδώ μια τροπολογία να το αλλάξουμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε να πάρει το λόγο από τους συναδέλφους. Ε, κανείς. Ωραία. Να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του. Κύριος Ερητέ. if I'm... Oui, euh, merci beaucoup pour... Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις τροπολογίες που ενεκρίθησαν επί του προϋπολογισμού ως προς το σχέδιο γνωμοδότησης. Εγώ είμαι υπεύθυνο ε, ε, της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, Παιδείας και Πολιτισμού. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με αυτές τις τροπολογίες, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι η Επιτροπή Πολιτισμού αποκατέστησε το αρχικό ποσό σε μια σειρά γραμμών, ιδιαίτερα ως προς τις, ε, τα εκτελεστικά γραφεία ΙΠΑ και Καναδά. Θα υπάρξει και συμπληρωματικός προϋπολογισμός για τις τρεις αυτές δράσεις. Σε σχέση με το πιλωτικό σχέδιο, για την πολιτιστική κληρονομιά. Εδώ πρόκειται για ένα πιλωτικό σχέδιο το οποίο θα μας απασχολήσει με τους ε, συναδέλφους που είναι υπεύθυνοι για θέματα δικαιοσύνης. Κινούνται παρόμοιες δράσεις, αλλά είναι ένας τομέας που δεν γνωρίζουμε πολύ καλά. Γι' αυτό θα έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους, αλλά είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε σχέση με τον προπολογισμό επικοινωνίας θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή γιατί πρότεινε την αποκατάσταση του αρχικού ποσού καθώς και τα επιπρόσθετα ποσά για να υποστηρίξετε την επικοινωνιακή μας πολιτική. Η Επιτροπή κυρία Βάλστραμ θα παρευρεθούν εδώ για να συζητήσουμε τι έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια ως προς την επικοινωνιακή μας πολιτική. Ο Κλάους Χέρνσεν, ο γενικός μας διευθυντής, ε, θα ήθελε να παρευρεθεί εδώ σε μία από τις επερχόμενες συνεδριάσεις για να συζητήσετε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την συνεργασία μας στον τομέα της επικοινωνιακής μας πολιτικής και με την ευκαιρία αυτή θα απαντήσει και τυχόν ερωτήσεις σας σε σχέση με επιμέρους στοιχεία του προϋπολογισμού. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε το λόγο. Όχι. Υπάρχουν συνάδελφοι που θα ήθελαν να θίξουν κάποιο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην Χέλγα. Φαίνεται πως όχι. Ε, προθεσμία λοιπόν για την καταβολή τροπολογιών για αυτήν την σύντομη γνωμοδότηση στη σελίδα 3 εδώ τον ε, εννοεί δηλαδή στο, υπό το σημείο 7 των εγγράφων σας το έχετε μπροστά σας το στέμαρτα 11 λοιπόν Σεπτεμβρίου την ερχόμενη εβδομάδα στις 12 η ώρα είναι η εκπνοή της ε, τις ε, προθεσμίες για την κατάσταση των τροπολογιών. Αν λοιπόν θεωρείτε πως μπορείτε να υποβάλλετε κάποια χρήσιμη τροπολογία έως τις 11 Σεπτεμβρίου, διαβιβάστε σας παρακαλώ τις τροπολογίες σας στην ε, γραμματεία. Η ψηφοφορία προφανώς θα λάβει χώρα στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου, δηλαδή 5 και 6 Οκτωβρίου. Εντάξει, έχουμε προχωρήσει λίγο ταχύτερα από ό,τι νομίζαμε. Ε, κυρία Βάλστρομ δεν είναι ακόμα εδώ αν μπορείτε να ειδοποιήσετε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ωραία. Αναβάλουμε λοιπόν μέχρι να είναι εδώ η κυρία Βάλστον το σημείο 8 και περνάμε στο σημείο 9 της μέρης σας διάταξης. Έγκριση δηλαδή των αποφάσεων των συντονιστών που συνεδρίασαν χθε το απόγευμα. Πάντοτε σας ε, διαβιβάζονται α, αυτές οι αποφάσεις των συντονιστών ε, το ίδιο βράδυ μέσω email. Δεν ξέρω αν έχετε ρίξει μια ματιά. Αλλά πάντα σας συνιστώ όταν θα έρχεστε για την δεύτερη μέρα των συνεδριάσεών μας ε, να ρίχνετε μια ματιά την προηγούμενη μέρα ή το πρωί στο email σας ε, για να ε, μπορείτε να ρίχνετε μια ματιά σε ό,τι αφορά τα αποτέλεσμα των, ε, τις αποφάσεις που έχουμε λάβει. Πάντως νομίζω πως υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους πράσινους και τους αριστερούς δηλαδή μεταξύ των πρασίνων και της αριστεράς σε ό,τι αφορά ε, την, ε, την ε, μία γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να αναλυθεί από κάποιον. Τι θέλετε να πει, κυρία Βέγκα. Ναι. Νομίζω ότι αν μου το επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, χτες προχωρήσαμε πολύ γρήγορα και ζητήσαμε αν μπορούμε να έχουμε μια μικρή προθεσμία σχετικά με την ανάθεση αυτής της έκθεσης για να μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Αυτό ήταν το αίτημά μας, αν μπορούμε να σας δώσουμε τη Δευτέρα το αργότερο μια απάντηση για να σας πούμε τελικά τι θα γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχαμε την αίσθηση ότι είχατε συμφωνήσει, αλλά πρόκειται να συμφωνήσετε. Ωραία. Sustainable Development, βιώσιμη ανάπτυξη λοιπόν. Πρόκειται για γνωμοδότηση και τη Δευτέρα θα μπορούμε να σας πούμε αν τελικά θα αναλάβει τη σύνταξη της ενόγω λόγω ε, η πράσινη πολιτική ομάδα ή η αριστερά. Κατά τα λοιπά θα ήθελα να ζητήσω την έγκρισή σας ε, των ε, πρακτικών των αποφάσεων των συντονιστών Λυπούμε λοιπόν, αν δεν διαβάσατε αυτέ τι ε, αποφάσει, αλλά σίγουρα θα το κάνανε οι βοηθοί σα και σα διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχει κάτι λανθασμένο. Μπορώ να λάβω την έγκρισή σα. Ποιο θέλει να πάρει το λόγο, κύριο Μάρτιν. Ζητώ συγγνώμη που θα πρέπει να πάρω πολύ σύντομα το λόγο. Γνωρίζω. Γνωρίζετε ότι εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον τρόπο που χειριστήκατε τα ζητήματα χθε, αλλά δυστυχώ ε, βάσει και τη συμβουλή που έχω πάρει από την ε, νομική υπηρεσία, καθώ. η η Northern Alliance δεν συμμετείχε σε αυτήν την ε, συζήτηση, ενδεχομένως ε, θα πρέπει να ε, αναφέρω εδώ αυτή την αμφιβολία μου και ενδεχομένως ότι αν υπάρξει κάποια, κάποιο πρόβλημα μελλοντικά ενδεχομένως να πρέπει να θεωρηθούν άκυρα αυτά τα αποτελέσματα, δηλαδή αυτές τις αποφάσεις γιατί δεν συμμετείχε η Βορειά Συμμαχία, η Northern Alliance. Ευχαριστώ, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε σχέση με αυτό. Παρακαλώ ακούστε με, είναι σημαντικά αυτά που λέμε εδώ. Ο κύριος Μάρτιν μας είπε ότι αποφασίσαμε σύμφωνα με την δική μας, ε, με το δικό μας καταστατικό ε, δεν μπορούμε να έχουμε συντονιστές, δηλαδή άτομα το μη εγγεγραμμένο να συμμετέχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών μας γιατί αναφέρεται στο καταστατικό ότι μόνο εκπρόσωποι πολιτικών ομάδων μπορούν να είναι συντονιστές, ε, πολιτικές ομάδες λοιπόν ορίζονται, ορίζουν συντονιστή που συμμετέχει. Ε, Όμω τελικά μετά από συζήτηση που κάναμε αποφασίσαμε ότι ο κ. Μάρτιν θα μπορεί να συμμετέχει υπό το καθεστώ παρατηρητή στη συνεδρίαση των συντονιστών. Και στην επόμενη ε, διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στην οποία εγώ έχω την Προεδρία, θα θέσω αυτό το ζήτημα ως επίγον σημείο στην ημερήσια διάταξή μας και θα συμφωνήσουμε λοιπόν σε εκείνη την ε, συνεδρίαση των Προέδρων των Επιτροπών τι θα κάνουμε με αυτό το ζήτημα. Και ο κύριος Μάρτιν τώρα μας ανακοίνωσε πως ε, εάν τα πράγματα παραμείνουν έτσι στο καταστατικό μας θα πάνε οι μη εγγεγραμμένοι έως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο και δικαιωθούν ε, τότε θα πρέπει να θεωρηθούν όλε οι αποφάσει που θα έχει λάβει μέχρι τότε η Επιτροπή μα άκυρε, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μα απασχολήσει, α μην φοβόμαστε, γιατί έτσι κι αλλιώ ακριβώ οι ίδιε θα ήταν οι αποφάσει αφού, αφού η πλειοψηφία συμφωνεί. Εν πάση περιπτώσει, α μην δημιουργούμε δυσκολίε, έτσι. Ε, υπάρχουν κάποιε δυσκολίε όπω και άλλε επιτροπέ. Άρα λοιπόν χαλαρά ήρεμοι θα αναμείνουμε λοιπόν τις αποφάσεις που θα ληφθούν, ενδεχομένως και αν εκδοθεί απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα αποδεχθούμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, όποια και αν είναι, ε, και μπορούμε να θα λάβουμε τις ίδιες αποφάσεις σε εκείνη την περίπτωση με αυτές που έχουμε λάβει. Κλείνω εδώ αυτό το ζήτημα, όχι περαιτέρω συζήτηση. Ε, περάσουμε στο σημείο τώρα ε, για τη συζήτηση με την κυρία Βάλστρομ, αλλά πρωτού το κάνουμε, εάν, θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχει κάποιο να δείξει κάτι υπό τα διάφορα αλλά όχι πια για αυτό το ζήτημα, κύριε Μάρτιν. Έτσι είπα ότι δεν θα συνεχιστεί η συζήτηση για αυτό το θέμα. Δεν θέλετε να θέσετε κάτι άλλο. Όχι τότε. Δεν σας δίνω το λόγο. Κυρία Χάνεμπα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για το θέμα 9 σχετικά με τις αποφάσεις. Ε, μπορούμε να το αναβάλουμε αυτό, διότι ακόμα έχω συζητήσεις με άλλους ε, συντονιστές. Νομίζετε ότι θα μπορούσαμε την έγκριση αυτή να την αναβάλουμε. Θέλει να πει κανείς κάτι σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Να κάνω λίγο για το... Yeah, yeah. Okay. Also wir werden die... Helga, möchtest du? Ελγκά, θέλεις να πεις κάτι για άλλο ζήτημα. Απαντάει η κυρία Τρούπελ. Ωραία. Να πάρουμε σοβαρά υπόψη μας αυτή την, αυτό το αίτημα της κυρία Σάνουμπα. Οπότε στην επόμενη συνεδρίασή μα τον Οκτώβριο θα ασχοληθούμε με αυτέ τι αποφάσει των συντονιστών, αλλά θα συνεχίσουμε τι εργασίε μα με βάση εκείνε τι αποφάσει που λήφθηκαν. Έτσι, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Έτσι, ωραία, αλλά μετά εκ νέου, α το πούμε έτσι, απόφαση επίσημη στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου για τι αποφάσει των συντονιστών. Κυρία Χάνιμπαλ, δεν είναι μόνο ότι ε, είναι το θέμα ε, των εκθέσεων. Πρέπει να ορίσουμε επίσης τα μέλη και αυτό είναι κατεπήγον. Σας παρακαλώ. Είναι 10 ε, παρατέταρτο. Μήπως μπορείτε να συντονιστείτε με τους άλλους μέχρι το τέλος της ημέρας, μέχρι το τέλος της συνεδρίασής μας μάλλον καλύτερα. Μαρία. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό να αρχίσουμε με αυτή την σπουδή που είναι ο ρυθμός που είχε επιβάλει η κυρία Πακ. Αλλά σε αυτή την περίπτωση από τα πρακτικά των συντονιστών, εγώ δεν μιλάω για μένα γιατί εγώ έχω τα πρακτικά, αλλά εν πάση περιπτώσει μιλήσατε για το ηλεκτρονικό ταχυδρόμιο. Πρέπει να εγκρίνουμε κάτι που αν ρωτήσετε την πλειοψηφία των μελών ούτε καν το έχει διαβάσει. Θα σας πρότεινα λοιπόν σήμερα να ανακοινώσετε ότι πριν από κάθε συνεδρίασή μας να κοιτάμε το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, ε, σήμερα όμως ε, ας πάρουμε μία ανάσα, ας το διαβάσουμε και να μπορέσουμε να το σχολιάσουμε, διότι δεν έχουμε πάρει τον ταχύτατο ρυθμό που είχε επιβάλει η κυρία Πάκα ακόμα. yeah. end of today. So, wir haben gestern Abend eigentlich in den meisten Bereichen. Ε, χθες ε, δεν είχαμε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο τομέα. Οπότε θα ήθελα να μας πει, κυρία Χάνιμπον, ποιοι είναι εκείνοι οι τομείς στους οποίους θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε περαιτέρω. Τότε θα πω ότι θα ψηφίσουμε, ότι θα συμφωνήσουμε δηλαδή, για όλα τα υπόλοιπα σημεία. Πείτε μας, κυρία Χάνεμπο, λοιπόν, ποια είναι τα σημεία που σας προβληματίζουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Βεβαίως. Πρόκειται για την κατανομή εκθέσεων. Για ποια μιλάτε, για ποια έκθεση μιλάτε. Δεν μπορούμε να αρχίσουμε με το ίδιο. Αυτό που, που κάναμε χτες. Ποια έκθεση νομοθετικού περιεχομένου διακόπτεται από την Πρόεδρο χωρίς μικρόφωνο και οι δύο ομιλήτριες. Ναι, μιλάμε για τις σεξουαλικές καταχρήσεις και την πορνογραφία. Ναι, μιλάτε για την πορνογραφία. Ως προς το voluntary report θα ανατεθεί μόνο τον Οκτώβριο την έκθεση για το έτος του εθελοντισμού. Μπορούμε να αποκλείσουμε αυτή την έκθεση υπαριθμών 9. να την κρατήσουμε κατά μέρος και να ψηφίσουμε για όλες τις υπόλοιπες. Και οι άλλοι ποια ήταν, Οι 9 και 11, γιατί οι πράσινοι και η αριστερά δεν ξέρουν πού, σε ποιο να τις αναθέσουν. Λοιπόν, 9 και 11 που βάζουμε κατά μέρος θα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο αυτές τις δύο εκθέσεις και για τις υπόλοιπες θα ψηφίσουμε. Νομίζω ότι ε, σήμερα και για τα σημεία 9 και 11 εάν μπορούμε μέσα στη συνεδρίαση Εάν ε, συμφωνήσουμε με τους συναδέλφους μπορούμε να επιλύσουμε το ζήτημα. Νομίζω κατά τη διάρκεια του πρωινού, έτσι ώστε να κλείσουμε αυτό το ζήτημα χωρίς να το αναβάλουμε για τον Οκτώβριο. Yeah. Κύριος Μάρτιν. Ναι, εγώ θα ήθελα να πάρω το λόγο για κάτι τελώς διαφορετικό. Αλλά κύριε Πάκη, σας παρακαλώ, μην μου θυμώσετε. Ε, ε, δεν με έχετε αντιληφθεί σωστά. Εγώ επικοδομητικός προσπαθώ να είμαι. Δηλαδή και εσείς θα ε, παλεύατε για τα δικά σας δικαιώματα και εγώ αναφέρομαι εδώ σε θεμελιώδη δικαιώματα των βουλευτών. Έχουμε περάσει τώρα στο σημείο υπό τα διάφορα και είχα αντιληφθεί ε, ότι έκλεισε η συζήτηση ε, για, το, για τις αποφάσεις των συντονιστών. Σας παρακαλώ μην μου θυμώνετε. Μην μου θυμώνετε και για μένα είναι πολύ δυσάρεστη αυτή η κατάσταση και θέλω πραγματικά να φτάσουμε το ταχύτερο δυνατό σε μια σύμφωνη γνώμη, σε μια συνένεση. Αλλά σας λέω ότι τα όσα συμβαίνουν εδώ ε, στο πλαίσιο των αποφάσεων των συντονιστών ε, ε, μερικές φορές δεν αντιλα... γίνονται αντιληπτά από τους υπόλοιπους. Οπότε σας λέω, ε, χωρίς να μου θυμώνετε και με συνενετικό πνεύμα, στο πλαίσιο της δημοκρατικής λήψης αποφάσεων, ε, σας ρωτώ, Είμαστε στο 8, είμαστε στο 9 που είμαστε. Ναι, ε, ξαναγυρίσαμε σε αυτό γιατί... Ε, η κυρία Χάνεμπα ζήτησε να παρέλθουμε σε αυτό. Ε, λέει ο κύριος Μάρτιν ότι σας λέω από νομική άποψη ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Απαντάει η κυρία Πακ, εντάξει σας ακούσαμε, βλέπετε τι είναι το 9. 9 λέει εδώ έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Ποτέ δεν είχα αντιμετωπίσει τόσες, ε, τόσα προβλήματα σε ό,τι αφορά την έγκριση των πρακτικών ή των αποφάσεων. Εν πάση περιπτώσει. Τι να κάνουμε, να, ακούσουμε τη, να, να, ακολουθήσουμε την πρόταση που έκανε ο κύριο Κουρέα. Δηλαδή, αφού έχουμε λίγο ακόμα χρόνο στη διάθεσή μα, γιατί είναι εδώ κυρία Βάτα, θέλουμε να το συζητήσουμε έξω από την αίθουσα. Στο σημείο 9 θα ήθελα να πω ότι η πρότασή σα με ικανοποιεί. Να εγκρίνουμε τα πρακτικά εκτό τα υποσυζήτηση σημεία Νομίζω ότι είναι ισορροπημένη πρόταση και έχω να υποβάλω και μία άλλη γιατί μας ζητήσατε να λάβουμε θέση επί πρακτικών που δεν διάβασα εγώ, δεν ήξερα ότι είναι στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομή. Άρα όταν ε, δουλεύουμε έτσι δεν είναι καλύτερα να γίνεται διανομή των πρακτικών το πρωί όταν έχουμε μία διημερίδα, στο το πούμε. Ναι, ήταν δικό μας το λάθος, γιατί έπρεπε να σας πούμε ότι στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο υπάρχουν τα πρακτικά. Για μία φορά το δέχομαι, τη δεύτερη φορά, την επόμενη δεν θα το δεχτώ. Διαβάστε το, ένας το διαβάσει κάποιος άλλος, δεν ξέρω ποιος το διαβάζει στη δική σας θέση. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Σκουρία είπε να αφήσουμε τα δύο σημεία κατά μέρο, το 9 και το 11, θα μας απασχολήσουν στην ε, επόμενη συνάντηση συντονιστών, αλλά θα έρθετε σε επαφή με τον κύριο Σκουρία και άλλους, αλλά θα ψηφίσουμε τα πρακτικά χωρίς το 9 και 11. Ποιοι είναι υπέρ των πρακτικών χωρίς τα σημεία 9 και 11. Ποιοι τάσσονται υπέρ. Κατά. κατά. Ευχαριστώ. Στο σημείο τώρα της κυρία Έλγα Τρούπελ. Είμαστε από τα διάφορα κύριε Μάρτιν, έτσι. Λοιπόν, κυρία Τρούπελ. Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των εργατησιών μας, θα ήθελα να ρωτήσω και νομίζω πως είναι και καινούριο. Ε, και για τους καινούριου συναδέλφους σε ενδιαφέρον το τι θα κάνουμε αυτό το έτος ε, ε, σε σχέση με το βραβείο Lux. Αυτό που κάνουμε είναι να διαλέξουμε ένα ε, έργο, κινηματογραφικό δηλαδή, από τα τρία τα οποία προβάλλονται εδώ και μετά αποδίδει ο κάθε βουλευτής κάποιους πόντους ε, και εκείνο τελικά η ταινία, δηλαδή το κινηματογραφικό έργο το οποίο θα κερδίσει ε, λαμβάνει δωρεάν υπότιτλους σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε επειδή είναι και φέτος ε, τρέχει αυτό το πρόγραμμα θα θέλαμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες γιατί θα θέλαμε αυτό να, να υπάρχει και μια προβολή όλης αυτής της πρωτοβουλίας και προς τα έξω. Ναι, ναι, θα επανέλθουμε σε αυτό, λέει η κυρία Πάκου, κύριο Μάρτιν. Ναι, ε, και εγώ το θεωρώ πολύ ε, ενδιαφέρον αυτό το ζήτημα. Ε, πέρσι α, ε, υπήρξε ένα ε, πολύ μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και σε ό,τι αφορά και τη ψήφιση και νομίζω πως το βραβείο θα πρέπει να έχει πιο σαφή ε, σύστημα ως προς το πώς ακριβώς αποδίδεται το βραβείο. Και σε αυτό συμφωνώ με την κυρία Τρούπελ. Ε, πάντως, ε, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα έχετε καθόλου κατά νου ποιε θα είναι οι ημερομηνίε συνεδρία τη Επιτροπή Πολιτισμού για, το, για του χρόνου, για να μπορούμε λίγο πολύ να προγραμματίσουμε Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιο άλλο. Όχι, λοιπόν, να πω λοιπόν κάποια πράγματα. Για του νέου συναδέλφου, λοιπόν, να επαναλάβουμε τι έχει γίνει εδώ. Αποφασίσαμε πριν από δύο χρόνια να ξεκινήσουμε την απονομή ενό βραβείου, ε, ούτω ώστε να προβάλλουμε λίγο περισσότερο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά το χώρο του κινηματογράφου και προκειμένου να καταδείξουμε, όπω είπε και η Χέλμπα, ε, Χέλγα, να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές ταινίες να έχουν περισσότερη προβολή και γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε ε, ένα βραβείο το οποίο είναι ιδιαίτερο. Είναι ε, πολύ ξεχωριστό. Δεν υπάρχει χρηματικό ποσό ως βραβείο, αλλά δωρεάν υποτιτλισμός σε όλες τις 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προβληθεί παντού. Αυτό είναι το, το ιδιαίτερο, αν θέλετε, το ξεχωριστό του στοιχείο αυτού του βραβείου. Η κριτική μας επιτροπή Ε, συντάσσεται από την υπηρεσία εικόνα ήχου, δηλαδή εικόνα ήχου, audio visual, δηλαδή άτομα από την αντίστοιχη μηχανία, μουσική και κινηματογράφου. Είχαμε λοιπόν μια προεπιλογή τριών έργων, τριών ταινιών πριν από το καλοκαίρι και ε, μετά Δευτέρα 2 Νοεμβρίου ε, θα έχουμε την προβολή μετά πάντα το μεσημέρι και το βράδυ Έχουμε δημιουργήσει δηλαδή μια κινηματογραφική αίθουσα στο, στον τρίτο όροφο πίσω από το Watchbox και όλοι οι ερετοί ευρωβουλευτές θεωρούνται μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Ρίξτε μια ματιά στις ταινίες. Εντάξει, θα πρέπει να θυσιάσετε κάποιο μεσημεριανό σας διάλειμμα ή ένα βράδυ και να αποφασίσετε από αυτές τις τρεις ταινίες που προβάλλονται εκεί, θα προβάλλονται για τις 14 μέρες, ποια προτιμάτε. Και θα μπορούμε να αποφασίσουμε και μέσω διαδικτύου. Το έργο λοιπόν εκείνο το οποίο θα επιλεγεί θα λάβει σε μια σύντομη εορταστική εκδήλωση κατά την Ορομέλεια το βραβείο. Θα έχουν προσκληθεί προφανώς ε, παραγωγική σκηνοθέτης, ε, ηθοποιή και ούτω καθεξής. Άννα Σιγκούλα, ε, και ο πολύ ε, γνωστός ε, Πορτογάλος σκηνοθέτης είχε έρθει κατά την τελευταία απονομή του βραβείου ένας πολύ σημαντικός Πορτογάλος σκηνοθέτης παραξελώς ε, έτσι είχαμε λοιπόν εκεί την προβολή και την απονομή του βραβείου στον νικητή είμαστε λοιπόν η κριτική επιτροπή εδώ είμαστε πάντα λοιπόν περισσότεροι πάντα περισσότερα μέλη στην Κρητική Επιτροπή από ό,τι για παράδειγμα για το Ρεβέο Καν, που είναι 25 μέλη Κρητική Επιτροπή. Θα ήθελα λοιπόν να σα ζητήσω, δεν το κάνουν όλοι, αλλά σα παρακαλώ κάντε το. Ε, είναι χαρά δηλαδή να δείτε αυτό το έργο, αυτή την ταινία ή αυτές τις ταινίες και μετά να μας δώσετε τη γνώμη σας. Εμείς είμαστε συνδιοργανωτές Επιτροπή ε, Πολιτισμού και Παιδείας. Εμείς δηλαδή μαζί με την ε, αρμόδια υπηρεσία audiovisual του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω πως έχει... Ναι, έχουμε προγραμματίσει ένα σοάρε, το βράδυ δηλαδή πριν από την ημέρα απονομής του βραβείου. Και ε, εκεί θα γίνει μια συζήτηση γιατί στο παρελθόν είχαμε προβλέψει διήμερο συζήτησης πριν από την απονομή που θεωρήσαμε πως είναι λίγο υπερβολικό οπότε ε, μέσα στο πλαίσιο αυτού του ΣΟΑΡΑ αποφασίσαμε τώρα να γίνει μια συζήτηση για αυτό το ζήτημα δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εδώ από την υπηρεσία audiovisual ε, αυτή τη στιγμή εδώ όχι θα ζητήσουμε πάντως επόμενη συνεδρίαση να προσέλθει εδώ μία, α, ε, κάποιος εκπρόσωπος από την πλευρά του Audiovisual και εμείς θα πάμε και στη Βιενάλε, θα είμαστε στις σκάνες Θα πάμε λοιπόν στην Βιενάλε και α, κατά συνέπεια θα προσπαθήσουμε και εκεί να προβάλλουμε το εν λόγω βραβείο. Οπότε όποιος ε, συνάδελφος έχει επαφή με κάποια από τα φοιτών, δηλαδή τα ένθετα των εφημερίδων για τις τέχνες, θα ήθελα να προβεί αντίστοιχε ενέργειε, να κάνει κάποια διαβήμιση, κάποια προβολή, ούτω ώστε να μην γίνεται μόνο γνωστή για τα χημικά ή οτιδήποτε άλλο Ευρωπαϊκή Ένωση στου πολίτε, αλλά να γίνεται γνωστή και για τα όσα αποτελούν το, την ψυχή τη Ευρώπη και την εικόνα τη προ τα έξω. Οπότε σα παρακαλώ επικοινωνήστε λίγο προ τα έξω. Δεν μπορεί να τα κάνει Επιτροπή. Μπορεί να προσπαθήσει η Επιτροπή και κάνει κάποιε δράσει, αλλά δεν θα εισακουστεί με τον ίδιο τρόπο που σα ακούνε εσά οι δικοί σα ε, άνθρωποι. Οπότε ε, κάντε κάτι, προβάλλετε όσο μπορείτε αυτό το βραβείο Λουξ, το οποίο άλλωστε θα συμμετέχετε και εσεί ω μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Πιο πολλά δεν μπορούσα να σας πω. Πάντως σας λέω, από τις 2 Νοεμβρίου για 14 ημέρες θα προβάλλετε μεσημέρι και βράδυ, θα προβάλλονται αυτές οι ταινίε. κάντε το κόπο, δείτε τις. Νομίζω είναι κάτι ωραίο. Κάτι το οποίο μα ε, εξοραίζει και εμά ω Επιτροπή και μα είπε άλλωστε και ο κλάδο του κινηματογράφου ότι κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει στο παρελθόν, είναι κάτι το καινούριο, α το προωθήσουμε. Κύριε Μάρτιν, έχετε το λόγο. Ε, κύριε Απάκ, είναι πολύ καλό αυτό, πολύ θετικό. Ε, ένα ακόμα ζήτημα θα ήθελα να πω. Ε, επιλέγουμε κάποιους οι οποίοι θα έρθουν εδώ, έτσι, σαν... Ε, ποιος τους επιλέγει, Κύριε Απάκ. Ναι, εμείς από κοινού με την υπηρεσία audiovisual ε, διαμορφώνουμε από κοινού δηλαδή τους προσκεκλημένους εκείνες τις προηγούμενες ημέρες του Σουαρέ δηλαδή. Ποιος, ποια είναι η αρμόδια επιτροπή, ρωτάει ο κύριος Μάρτιν. Συνεργαζόμαστε. Συνεργαζόμαστε, αλλά βασικός διοργανωτής είναι η υπηρεσία audiovisual του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα, έτσι. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η υπηρεσία για να αναλαμβάνει τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά σας λέω πάντα σε συνεννόηση μαζί μας και το γεγονός ότι η πρόεδρος ε, της Επιτροπής μπορεί να παρουσιάζει αυτό το βραβείο ε, στην Biennale σημαίνει ότι δεν μας ε, παρακάμπτουν αλλά ότι συμμετέχουμε ενεργά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλή σας μέρα και πάλι. Ε, για να φτάσουν αυτά τα, τα τρία φιλμ στην α, Κριτική Επιτροπή που είμαστε εμείς και όλοι οι άλλοι ενεργοί βουλευτές ε, προκύπτει κάποια υπάρχει κάποια προκήρυξη ε, πρόσκληση για να υποβληθούν ή κάποιο τα επιλέγει. Ευχαριστώ. So, diese Filme kommen nicht in den Ausschuss. Όχι, δεν διαβιβάζονται στην Επιτροπή μας αυτές τις ταινίες. Έχουν προεπιλεγεί τρεις ταινίες και από τις 2 Νοεμβρίου και μετά προβάλλονται σε αυτήν την κινηματογραφική αίθουσα που υπάρχει πίσω από τη Watchbox στον τρίτο όροφο. Θα μπορεί δηλαδή όλο το κοινοβούλιο να, να, να βλέπει αυτό το ταινίο. Δηλαδή υπάρχουν, θα υπάρχουν μεγάλε αφήσει εκεί σε όλο το κοινοβούλιο που θα ενημερώνουν. Ρίξτε μια ματιά, αλλά ναι, θα λάβετε από εμά και μια έγγραφη ενημέρωση ω προ το πότε θα αρχίσει η προβολή, πόσο θα διαρκέσει, οι ημερομηνίε ε, συγκεκριμένα που θα προβάλλονται αυτές οι ταινίες και με βάση αυτή την ενημέρωση θα μπορείτε να αποφασίσετε. διάλεξε αυτά τα τρία τη τρεις ταινία, γιατί δεν έχουμε δέκα. Αυτή ήταν η ερώτησή μου. Ε, δέκα ταινίε είχαν προταθεί. Δέκα ταινίε. Και από αυτές τις δέκα ταινίε υπάρχουν ταινίε. έτσι, όχι αυτές που έχουν ήδη προβληθεί στον κινηματογράφο, εξετάστηκαν από μια κριτική επιτροπή και αυτές προεπέλεξαν τρεις που θεώρησαν ότι ε, ανταποκρίνονταν περισσότερο στο ευρωπαϊκό πνεύμα. Και εμείς θα αποφασίσουμε τώρα, θα επιλέξουμε από τις τρεις αυτές τις ταινίες που έχουν γίνει μία. Ε, συνάδελφε. Ε, κυρία Πρόεδρε, γνωρίζετε ότι είμαι νέα συνάδελφο. Ε, δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώ τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με αυτό το βραβείο. Δηλαδή, θα μπορούμε να δούμε αυτέ τι ταινίε μόνο στην κινηματογραφική αίθουσα. Γιατί ε, ήταν πάρα πολλοί οι οποίοι είχαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έβλεπαν δηλαδή το, ε, αυτές τις ταινίες οπότε θα ήθελα να ρωτήσω μήπως θα ήταν δυνατό να προβάλλονται και στις ε, τηλεοράσεις που έχουν στα γραφεία τους οι ε, βουλευτές αυτές τις ταινίες ώστε να μπορούν να, βλέπουν, να δουν αυτή, την, ε, αυτές τις ταινίες. Εγώ είμαι πολύ υπέρ λέει η κυρία Πακ των νέων μέσων αλλά ε, την ταινία πρέπει να τη βλέπουμε στον κινηματογράφο. Και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να δει μια ταινία ενώ γράφει ταυτόχρονα και κάτι μια σημείωση. Δηλαδή, όλοι νομίζω θα μπορούσαμε να, να... είναι και μια, μια πολύ ωραία εμπειρία να πάμε στην κινηματογραφική αίθουσα και να δούμε τι ταινία. Και πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ ε, σε ποιον δεν θα άρεσε κάτι τέτοιο, δεν θα μπορείτε ούτε popcorn να αγοράσετε, ούτε chips εκεί. Το, το καλύτερο πράγμα, το πιο ωραίο πράγμα, το τέλειο. Θα, πάρε, θα λάβετε, σας λέω, εγκαίρως ε, τις ημερομηνίε, οπότε μπορείτε ακριβώ να οργανώσετε το χρόνο σας. Ε, άμα δηλαδή εμείς ως ε, Επιτροπή Πολιτισμού δεν μπορούμε να πούμε το χρόνο για να πάμε στην κινηματογραφική αίθουσα, ποιο θα το βρει το χρόνο. Α, όποιος δεν ξέρει να πηγαίνει ακόμα στον κινηματογράφο, ε, ήρθε η ώρα να το μάθει. Ωραία. Λοιπόν, και θα λάβετε και εγγράφος από εμάς τα όσα μπορείτε κι εσείς να διαβάσετε στους δικούς σας ε, πολίτες ε, εν ενημέρωσης. Καλώς κλείνουμε με αυτό το ζήτημα. Καλώς ορίζω εγκάρδια εδώ την κυρία Βάλστρομ μαζί μας, η αρμόδια επίτροπος για την επικοινωνία. Ε, έχουμε συζητήσει μαζί σας πάρα πολύ στο παρελθόν. Έχετε ακούσει πάρα πολλά από εμά, αλλά και βέβαια έχει δώσει και στη δική μας επιτροπή πάρα πολλά, γιατί και εκείνη βρίσκεται πολύ κοντά στους πολίτες, δεν είναι μια επίτροπη, επίτροπος η οποία βρίσκεται κάπου εκεί μακριά, στο δικό της βάθρο, αυτά μου είπαν και από τη Σουηδία. Και μπορείτε να μας πείτε τώρα τι θέλετε να κάνετε εσείς και τι αναμένετε και από εμά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με δεχθήκατε εδώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ που εξελέγετε ή επανεξελέγετε ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την επιλογή σας να συμμετάσχετε σε αυτήν την Επιτροπή που έχει ευρύ φάσμα σημαντικών αρμοδιοτήτων από την παιδεία στην πολιτική επικοινωνία. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε σε αυτό το πρώιμο στάδιο να έρθω στην Επιτροπή σας για να συζητήσουμε την πολιτική επικοινωνία και ε, τις ε, που θα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Είχα όπως είπε και η κυρία Πρόεδρος, εξαίρετη συνεργασία με την Επιτροπή σας κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών και οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες ξεκινήσαμε δεν ήταν εύκολες. Να τον αναπτύξουμε μια συνεκτική στρατηγική επικοινωνίας και αποτελεσματικά εργαλεία για καλύτερη επικοινωνία της Ευρώπης απαιτήσε πολιτική βούληση και δέσμευση ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαθέσουμε τα οικονομικά και ανθρώπινα ε, μέσα και πόρους και για να έχουμε αλλαγές στη θεσμική μας κουλτούρα αυτή η Επιτροπή υπήρξε ε, ισχυρός και πιστός ε, σύμμαχος. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην Doris Πακ, η οποία είναι πεπειραμένο μέλος αυτής της Επιτροπής ε, και της αξίζει αυτή η προεδρία αυτής ε, της Επιτροπής και να αναφερθώ και στην Helga Τρούπελ πρώτη αντιπρόεδρο αλλά βλέπω και πολλά νέα πρόσωπα εδώ σήμερα και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι πάντοτε ανοιχτή στις ιδέες σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας. Η συνεργασία, η εταιρική σχέση στην επικοινωνία είναι ουσιώδης όχι μόνο με την ευρία έννοια των θεσμών αλλά και προσωπικά. Η αρχή μιας νέας θητείας είναι βεβαίως μια καλή ευκαιρία για να κοιτάξουμε προς τα πίσω. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να σας μιλήσω λίγο για τις προσπάθειες των πέντε τελευταίων ετών για να μπορέσουμε εσείς και εγώ τελικά να εξαγάγουμε ορισμένα διδάγματα για το μέλλον της πολιτικής επικοινωνίας και να κάνουμε μερικές προτάσεις για το πώς εσείς ως βασικοί παίκτες στο Κοινοβούλιο σε αυτόν τον τομέα μπορείτε να εξασφαλίσετε οι μεταρρυθμίσεις που θα ξεκινήσουμε μαζί θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Και αυτό είναι χρήσιμο για τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου. Γυρίζουμε πίσω στο 2004 όταν η Επιτροπή Βαρόζο άρχισε να εργάζεται για πρώτη φορά με ε, το χαρτοφυλάκιο της επικοινωνίας, όχι μόνο με τον τύπο και την ανημέρωση. Άκουσα πολύ συχνά στις συζητήσεις ότι η επικοινωνία είναι μια αδύνατη, ανέφικτη αποστολή ε, ε, η, η προπαγάνδα γενικά το λέει αυτά, ότι η Ευρώπη βρίσκεται πολύ μακριά, είναι πολύ περίπλοκη για να εξηγηθεί σε τόσες πολλές γλώσσες ε, και υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες ε, που είναι με στο παιχνίδι και υπάρχουν πολλά συμφέροντα και πάντοτε απαντώ ότι εγώ δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτή την αποστολή, είναι πολύ ελκυστική στο, έχουμε την βελτιωμένη έκδοση της συνθήκης της Λισαβόνας. Πολλοί πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι περίπλοκη, αλλά και η ζωή είναι περίπλοκη. Δεν ξέρω ε, πώς, ε, τι γίνεται η, ε, η κυκλοφορία, ο φούρνος μικροκυμάτων πώς λειτουργεί, αλλά ξέρω ότι διευκολύνουν τη ε, ζωή μου. Εμεί προσπαθούμε τα άτομα να αγαπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό διάλογο με τους πολίτες και να δημιουργήσουμε μια συζήτηση πανευρωπαϊκή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να πλησιάσει τους πολίτες και έτσι να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στους πολίτες και σε αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένες λύσεις, ότι η Ευρώπη ε, είναι μια πρόκληση. Δεν είναι όμως μια αφηρημένη πολιτική, είναι κάτι το συγκεκριμένο και αφορά ε, τους λαούς. Η επικοινωνία λοιπόν στην Ευρώπη, της Ευρώπης, η προβολή της Ευρώπης ε, δεν είναι σαν να πουλάει κανείς ε, κάλτσες ή κινητά τηλέφωνα. Για μένα η επικοινωνία είναι απαραίτητο στοιχείο της δημοκρατίας και είναι δημοκρατικό δικαίωμα των πολιτών να ενημερώνονται για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις που θα τους επηρεάσουν για να μπορέσουν να δεσμευθούν, να συμμετέχουν και να έχουν μια φωνή. Η συμμετοχή στην πολιτική ζωή είναι αυτό που δίνει στην πολιτική μια νομιμότητα και έχω τονίσει το επιχείρημα τα πέντε τελευταία χρόνια ότι η επικοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί την δημοκρατία. Η συμμετοχική δημοκρατία, η ζωντανός διάλογος και η συζήτηση θα πρέπει να κινητοποιήσουν τους πολίτες να λάβουν μέρος στη διαδικασία της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Και αν μπορούν οι αποφάσεις να περάσουν τα σύνορα, αν μπορούν να περάσουν στο ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε Ασφαλώς πρέπει να προωθήσουμε μια διασυνοριακή συζήτηση. Τελικά το μέτρο της επιτυχίας είναι ε, πώς οι αποφάσεις αυτές έχουν σχέση με τις προσδοκίες ε, των λαών. Στην αρχή λοιπόν της θητείας μου επαναπροσδιορίσα τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ασχολείται με το θέμα αυτό, πώς περνάει από την ενημέρωση στην επικοινωνία, από τις Βρυξέλλες στον Πρνό από τους θεσμούς, τους πολίτες και από την ιστορία στο μέλλον. Επρόκειτο για τον εξυγχρονισμό ε, του δρόμου μιας λωρίδας ώστε να γίνει ένας δρόμος διπλής λωρίδας με ενεργό διάλογο με τους πολίτες. Αυτό συνεπάγεται πολιτιστική αλλαγή στην Επιτροπή. Εάν στο παρελθόν το βασικό κριτήριο επιτυχίας είναι να κάνουμε τα πρωτοσέλιδα του Financial Times ή της Le Monde σήμερα, το κριτήριο είναι να υπάρχει μια μεγάλη διαβούλευση δημόσια πριν από μια πρόταση που θα οδηγήσει σε μια πολιτική. Να υπάρξει επίσης μια γενική συζήτηση για το πώς οι πολίτες θέλουν να προχωρήσει η Ευρώπη πώς αισθάνονται οι πολίτες στην Ευρώπη και πώς μπορούν να την επηρεάσουν. Έχω προσδιορίσει τρεις αρχές στους, σαν ακρογωνιαίους λίθους της εργασίας μου. Να ακούμε καλύτερα τις ανησυχίες των πολιτών, να εξηγούμε στους πολίτες τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να κατεβαίνουμε στο τοπικό επίπεδο, ούτως ώστε οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επικοινωνώντας μαζί τους ε, στις δικές, στα δικά τους μέσα ενημέρωση στο τοπικό επίπεδο και επίσης έχουμε την πρωτοβουλία στα σχολεία. Οι αξιωματούχοι μιλούν στα σχολεία, στους μαθητές για την δουλειά τους, για την πείρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δίνει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια δυνατότερη ε, σχέση ε, με την Φινλανδία, με την Ιταλία, καλύτερη σχέση με τις Βρυξέλλες. Πρέπει λοιπόν τα ίδια τα θεσμικά όργανα να πηγαίνουν στα σχολεία με βάση τις αρχές αυτές και είχαμε ένα πρόγραμμα δράσης για να μεταρρυθμίσουμε την εσωτερική μας δομή, να εξυγχρονίσουμε και να κάνουμε πιο επαγγελματική την προσέγγιση μας και να αποκεντρώσουμε τη δομή μας. Έχουμε προτείνει 50 δράσεις που υλοποιήθηκαν επιτυχώς. Αυτό χρειαζόταν επαγγελματίες. Έπρεπε να τους στρατολογήσουμε, έπρεπε να αναγνωρίσουμε το ρόλο ε, του προσωπικού της Κομισιόν στην επικοινωνία. Θα έπρεπε να έχουμε περιλήψεις αναγνώσιμες ε, για όλους τους πολίτες μας σχετικά με τις νομοθετικές μας προτάσεις. Μπορώ να σας δώσω μερικά παραδείγματα από εφ' εξής, όλες οι προτάσεις που στέλνουμε στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, πρέπει να έχουν μια περίληψη μονοσέλιδη για τους πολίτες που να εξηγεί σαφώς στους πολίτες περί τίνος πρόκειται. Επίσης, σημαντικό μέρος αυτού του εξυγχρονισμού ήταν στον τομέα των οπτικοακουστικών ακόμα ε, και στο διαδίκτυο. Στόχος της επικοινωνίας ε, ήταν ε, με βάση ε, την χρησιμοποίηση των μέσων που προτιμούν οι πολίτες. Είδαμε ότι λιγότερο από 10% του χρόνου των ειδήσεων είναι αφιερωμένος σε ειδήσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν μεγαλύτερο μερίδιο. Ε, το διαδίκτυο και τα οπτικοακουστικά μέσα είναι ε, βασικά θέματα για την διεύρυνση της ε, στρατηγικής επικοινωνίας. Είχαμε να δικήσουμε τον ιστότοπο Europa και ήταν κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Ε, κάνουμε την πρόσβαση στην πύλη ευκολότερη ε, και ευκολότερη την πλοήγηση για ενημέρωση. Θέλουμε ε, να έχουμε επίσης και αλλού παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διαδίκτυο, στον, στην ιστοσελίδα YouTube, Tube που από τον Ιούνιο 2007 είναι μέρος της πύλης της δημοφιλούς YouTube που περιλαμβάνει τώρα πάνω από 230 βίντεο ήμουν ο πρώτος επίτροπος που είχα blog, τώρα είμαστε 7 και αυτό διευκολύνει τη συζήτηση σε 23 γλώσσες για διάφορα ευρωπαϊκά θέματα. Οι περισσότεροι πολίτες Ευρωπαίοι χρησιμοποιούν ακόμα την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για τις ειδήσει για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Γι' αυτό υιοθετήσαμε μια οπτικοακουστική στρατηγική που συνεπάγεται την ενθάρρυνση της δημιουργία ε, ενός δικτύου σταθμών ε, και έχουμε ακροατήριο που είναι 20 εκατομμύρια άτομα κάθε μέρα. Ε, στην, στο, έχουμε το RT Radio στο Βέλγιο, ε, και έχουμε τις ευρωπαϊκές ειδήσει ε, και σύντομα θα έχουμε ένα παρόμοιο δίκτυο τηλεοπτικών ε, σταθμών που θα απευθύνεται σε 40 έως 60 εκατομμύρια θεατές. Διπλασιάσαμε την, την ικανότητά μας σχετικά με την Europe by Satellite και με 400 κανάλια σε ολόκληρο τον κόσμο. Βεβαίως αυτό απαιτεί οικονομικά μέτα Χάρη στο Κοινοβούλιο μπορέσαμε να αυξήσουμε τους πόρους μας για την εργασία επικοινωνίας και ελπίζω ότι θα μπορώ να βασίζομαι σε εσά ούτως ώστε να αντισταθείτε σε κάθε προσπάθεια μείωσης του ε, μελλοντικού προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ. Ακόμα και με αυτές τις αυξήσεις, οι συνολικές δαπάνες για την επικοινωνία είναι 0,2% του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 40 λεπτά κατ' κατέτος και αυτό περιλαμβάνει την χρηματοδότηση 33 γραφείων ε, αντιπροσώπησης και δεν νομίζω ότι με τους περιορισμούς που έχουμε τα πράγματα θα αλλάξουν μέχρι το 2013. Βεβαίως, η επικοινωνία της Ευρώπης δεν είναι μόνο ευθύνη της Επιτροπής. Εναπόκειται στα εθνικές κυβερνήσεις, στα πολιτικά κόμματα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δράσουν επίσης. Έχουμε λάβει ορισμένα μέτρα για συνεργασία, εταιρικέ σχέσεις με ορισμένες ε, χώρες. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρώπη, στα σπίτια της Ευρώπης και τώρα έχουμε δημόσιους χώρους όπου το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει σεμινάρια, ε, διαλέξεις, ε, συζητήσεις και ελπίζω ότι θα συμμετέχετε, θα συμμετάσχετε σε αυτές τις δραστηριότητες. Αρχίσαμε με τρία κράτη-μέλη και ελπίζω ότι θα έχουμε 11 το επόμενο έτος. Και Επίσης, πέρσι δημιουργήσαμε λίγη ιστορία τον Οκτώβριο, διότι συμφωνήσαμε για μια πολιτική δήλωση που έχει ως τίτλο ε, «Επικοινωνία της Ευρώπης σε συνεργασία» που υπόγραψαν το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και η πρώτο-πρώτο ε, ε, θέμα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν οι εκλογές, οι ευρωεκλογές και νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή εργασία. Μερικοί λένε, μα βεβαίως, αλλά η συμμετοχή στις ευρωεκλογές δεν ήταν μεγάλη. Πού είναι λοιπόν η επιτυχία ότι σε 11 χώρες αυξήθηκε η συμμετοχή. Εκεί όπου χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονα μέσα όπως η ηλεκτρονική ψήφος αυξήθηκε η συμμετοχή και εκεί όπου υπό τα πολιτικά κόμματα έκαναν προεκλογική εκστρατεία για ευρωπαϊκά θέματα η συμμετοχή αυξήθηκε. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αλλαγή για το πώς αντιμετωπίζουμε τις ευρωπαϊκές υποθέσεις σε καθημερινή βάση. Είναι ευθύνη όλων των πολιτικών παραγόντων σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο να αρχίσουν συζητήσεις για ευρωπαϊκά θέματα όπως το κάνουν για εθνικά θέματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε οι πολίτες να ψηφίσουν για ευρωπαϊκά θέματα αν αυτά συζητούνται μόνο με μερικές εβδομάδες στην προεκλογική εκστρατεία. Πρέπει να επενδύσουμε σε πολιτικές προσπάθειες. Και έρχομαι ε, για τα στα διδάγματα. Τα τελευταία πέντε χρόνια αρχίσαμε λοιπόν αυτό το εγχείρημα, αλλά με τις προσπάθειές της θα αποφασιστεί αν το εγχείρημα αυτό θα συνεχιστεί. Έχω τρεις συγκεκριμένες ε, προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, από την δική μου την πείρα, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπάρξει επίτροπος που να είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά στην επόμενη Επιτροπή κάποιος που να μπορεί να επισύρει την προσοχή των συναδέλφων πάνω στα χιλιάδες θέματα που έχει στην ατζέντα της η Νομίζω ότι ο ρόλος αυτός θα ενισχυθεί αν η πολιτική επικοινωνία συνδεθεί με άλλες απόψεις της ηθαγένειας στην Κομισιόν, προγράμματα ηθαγένειας, δικαιώματα των πολιτών και η νέα πρωτοβουλία για την συνθήκη της Λισαβόνας αυτό θα είναι ένα σήμα, μια ένδειξη ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να παίρνει σοβαρά το θέμα αυτό. Δεύτερον, το κοινοβούλιο αυτό θα είναι υπεύθυνο για την επαναδιαπραγμάτευση του νέου πολιετούς χρηματοοικονομικού πλαισίου που θα αρχίσει το 2013. Αν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχετε συναπόφαση για τον προϋπολογισμό και το πλαίσιο αυτό θα απαιτήσει την συνένεσή σας. Συνεπώς θα έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε η ε, δημοσιονομική αρχιτεκτονική της Ένωσης να εξασφαλίσει τα, τους απαιτούμενους πόρους για την προώθηση του διαλόγου και της δέσμευσης των πολιτών. Ελπίζω λοιπόν ε, να διαφυλάξετε αυτούς τους πόρους για την επικοινωνία. Και τρίτον, αυτή η συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής και Συμβουλίου είναι κάτι το καινούριο, αλλά θα λειτουργήσει αποτελεσματικά αν όλα τα θεσμικά όργανα ε, προσπαθήσουν να συνεργαστούν. Υπάρχει ένα σώμα ε, που είναι το IGI, ε, το Διεθνής Ομάδα ε, διαθεσμική, η διαθεσμική με συγχωρείτε, ομάδα για την πληροφόρηση, όπου μαζί το Συμβούλιο, Επιτροπή και το Κοινοβούλιο προγραμματίζουν μαζί τις προτεραιότητες επικοινωνίας για το επόμενο χρόνο. Είναι λοιπόν συμφέρον μας όλοι μαζί να συνεργαστούμε και αν τεθεί σε ισχύ η νέα συνθήκη θα έχετε μια βάση για ισχυρότερη συνεργασία εις το μέλλον. Και τέλος, τέλος, αν μου το επιτρέπετε, ε, μία συμβουλή, διότι υπάρχουν πολλοί στην Ευρώπη που ακόμα πιστεύουν ότι δεν είναι έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχολείται με την επικοινωνία για ευρωπαϊκά θέματα. Ή τα δημοψηφίσματα ε, στην Γαλλία, στις κατοχώρες, στην Ιρλανδία. Μας έμαθαν κάτι, μας έμαθαν ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να παρτίζεται μόνο από ελίτ που λαμβάνουν αποφάσεις και κλεισμένων των θυρών. Πρέπει να πλησιάσουμε, να τίνουμε χείρα ε, στους πολίτες, να τους ενημερώνουμε για τις ευρωπαϊκές πολιτικές ε, και να, για να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε αυτόν τον τομέα εργασίας και να μην περιθεροποιήσουμε ε, ή γελιοποιήσουμε το θέμα αυτό, διότι το μέλλον της Ένωσής μας θα εξαρτηθεί από το πώς καλά ε, θα ε, επιτύχουμε όταν λαμβάνουμε αποφάσεις ε, να προέρχονται από τις επιθυμίες των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. σε όλα αυτά τα ζητήματα που θίξατε είμαστε σαφώς από την πλευρά της δικής μας Επιτροπής στο πλευρό σας. Βέβαια, για όλα όσα κάνετε πάντα θα υπάρχει κριτική. Από τη μία πλευρά κάποιοι λένε ότι κάνετε προπαγάνδα, κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν κάνετε πολλά. Πάντως ε, όλα όσα πρέπει να κάνετε δεν μπορείτε να τα καταφέρετε μόνοι σας. Και αν μόνο εσείς δραστηριοποιούσασταν εδώ δεν θα ήμασταν επιτυχείς. Χρειαζόμαστε και τις εθνικές κυβερνήσεις κατά τη διάρκεια των 5 ετών, που οποίοι θα πρέπει να κάνουν κάτι για να ευαισθητοποιούν τους πολίτες ε, ε, των δικών τους χωρών και ε, νομίζω πως μας αφορά όλους το να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η Ευρώπη λειτουργεί σωστά. Εν πάση περιπτώσει και όπως είπατε σωστά κυρία Επίτροπε δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα αλλά ό,τι γνωρίζουμε είναι προς όφελος μας. Πρέπει πάντως αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να μιλήσουμε στην καρδιά των ανθρώπων. Και πώ θα μιλήσουμε στην καρδιά των ανθρώπων μόνο αν είμαστε εκεί παρόντε, σε τοπικό επίπεδο. Γι' αυτό έχετε δίκιο όταν λέτε go local. Δραστηριοποιηθείτε δηλαδή στο τοπικό επίπεδο. Καλώ, έχουμε πολλού ομιλητέ που θέλουν να πάρουν το λόγο. Καταρχήν να δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, κυρία Χέλγα Τρούπελ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την εισήγησή σα και για τι προτάσει σα. Και θα ήθελα να πω ότι τάσσομαι υπέρ των συγκεκριμένων προτάσεών σας, διότι πιστεύω ότι είναι σημαντικό να έχουμε έναν επίτροπο ή μία επίτροπο για θέματα ε, ηθαγένειας ε, και επικοινωνίας, να κινηθούμε σε τοπικό επίπεδο και να δούμε τις ε, διαδικασίες του Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να τίνουμε χείρα προς τους Ευρωπαίους πολίτες, ιδιαίτερα με τα πολυμέσα, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την παιδεία, την εκπαίδευση, τα πολιετή προγράμματα, έτσι ώστε να τίνουμε αυτή την χείρα προς τους πολίτες στην καθημερινή του ζωή. Θα πρέπει λοιπόν να το καταστήσουμε αυτό απόλυτα σαφές και αφορά άμεσα την Επιτροπή μας. Έχετε απόλυτο δίκαιο ότι για όλα αυτά χρειαζόμαστε επαρκείς πόρους και βρισκόμαστε πολύ πίσω και εγώ δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη για τον προϋπολογισμό μας ε, για θέματα πολιτισμού και παιδείας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει πολλά. Υπάρχει η χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στους νέους, στην εκπαίδευση και στην έρευνα, καθώς και την επικοινωνία και τον πολιτισμό. Διαφορετικά δεν θα κερδίσουμε τους ανθρώπους. Ξέρω βεβαίως ότι είναι πολύ δύσκολο για τα κράτη-μέλη και τους Υπουργούς Οικονομίας και οικονομικών, αλλά με το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να επιμείνουμε. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και ελπίζω να φτάσουμε σε νέες πλειοψηφίες. Και το τρίτο σημείο είναι ότι τα τρία θεσμικά όργανα πρέπει να συνεργαστούν θα πρέπει να επικοινωνούμε, να ξέρουμε ποια είναι τα κοινά μας συμφέροντα, τα κοινά συμφέροντα, ακόμα κι αν υπάρχουν διαφωνίες και ρήξεις. Υπάρχει όμως ένας κοινό παρονομαστής ως προς τον σφαιρικό μας ρόλο, το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδοκινοτικά αλλά και προς τα έξω. Ποια είναι τα καθήκοντά μας και η ευθύνη μας στη διεθνή σκηνή. Θα ήθελα και το παραδέχομαι αυτό. Θα ήθελα να πω ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας αποφάνθηκε ως προς τη συνθήκη της Λισαβόνας. Βεβαίως ε, τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να καταστήσουν σαφές ότι η Ευρώπη αποτελεί αναφέρατο καθήκον τους και θα πρέπει να τίνουμε χείρα προς τους πολίτες αλλά το τελευταίο δημοψήφισμα στην Ιρλανδία μας έδειξε ότι έχουμε να κάνουμε με τους πολιτικούς ηθήνοντες και μια πολιτική ελίτ που θα πρέπει να συνεργαστεί. Μιλάμε για εθνική δημοκρατία και υπερεθνική δημοκρατία. Θα πρέπει να συνταχθούν αυτές οι δύο συνιστώσεις, δηλαδή οι πολιτικοί ηθήνοντες και η πολιτική ελίτ θα πρέπει να το προωθήσει αυτό και στα κράτη-μέλη, διότι η Ευρώπη ε, απαρτίζεται από τα κράτη-μέλη, από την πολιτική τάξη και τους ηθήνοντες και την ευρωπαϊκή σκηνή και τους πολίτες βέβαια. Τα τελευταία χρόνια στα κράτη-μέλη αυτή η πολιτική γνώση βρίσκεται πολύ πίσω. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε ότι η Ευρώπη αφορά μόνο εμάς. Χρειαζόμαστε περαιτέρω συζητήσεις. Είναι πολύ καλό που έχουμε μία επίτροπο που είναι υπεύθυνη για θέματα επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει προπαγάνδα, διότι μιλάμε για πληροφορίες και για το πόσο οι άνθρωποι μπορούν να συμμετέχουν στα δρόμενα. Δεν πρόκειται για μία μηχανή προπαγάνδας δηλαδή εδώ αποτελεί στο τμήμα μιας πολιτικής ε, συζήτησης και θα ήθελα να τονίσω και το τελευταίο. Εμείς ε, οι ευρωβουλευτές είμαστε πρέσβεις της Ευρώπης και θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές τις εκλογικές μας περιφέρειες ότι θα πρέπει να γίνουν επιτόπιες συζητήσεις γιατί εμείς είμαστε ο σύνδεσμος μεταξύ εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών. Είναι πολύ καλό να έχουμε μια επίτροπο, αλλά εμείς ως Ευρωβουλευτές δεν πρέπει να ξεχνάμε τα καθήκοντά μας, πού ζούμε και πώς πρέπει να δράσουμε ως σύνδεσμος. Κυρία Μπαντία, ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Βάλστρομ για την παρουσία της εδώ που γνωρίζουμε ήδη και την διεξοδική της παρουσίαση και τις πρωτοβουλίες της. Τις ε, συμμερίζομαι όλες. Θα ήθελα όμως να επιμείνω σε ένα ζήτημα το οποίο θίξατε και εσείς. Είπατε για τα ευρωπαϊκά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να μας απασχολήσουν σε καθημερινή βάση. Αυτό είναι το κλειδί για να φτάσουμε στους πολίτες, διότι μιλάμε για ε, ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Νομίζω ότι δεν, έχει, δεν είναι μια έννοια η οποία έχει ριζώσει στη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών. Θα πρέπει ο πολίτης να νιώσει ότι ανήκει κάπου και οι πολίτες μας δεν ε, νιώθουν ότι ανήκουν στην Ευρώπη. Επ' αυτού θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω το εξής. Είναι ίσως μία αιμονή μου, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλύτερα όλα τα εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέσα που διαθέτουμε, ιδιαίτερα την τηλεόραση, διότι αυτά τα πολυμέσα μπαίνουν στα σπίτια των ε, πολιτών. Όποιος ενδιαφέρεται μπαίνει στο διαδίκτυο, ψάχνει, ψάχνεται. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία έχει μόνο αυτό το μέσο, το μέσο που διαθέτει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή η τηλεόραση θα πρέπει να μιλάει για την Ευρώπη. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με τις περιφερειακές τηλεοράσεις και τα τοπικά δίκτυα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακίνου. Μακλάκιν, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο που βρέθηκε, παραβρέθηκε εδώ σήμερα. Συμφωνώ με την ενθάρρυνση της καθημερινής ε, ε, ζωηρής συζήτησης, έτσι ώστε να πάρουν μορφή τα θέματα αυτά μέσω της συζήτησης. Παρόλα αυτά, θεωρώ σήμερα ότι πολλές δράσεις ε, θεωρούν πρόκριμα την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρούν οι Ιρλανδοί ότι δεν έχει ληφθεί υπόψη η θέλησή τους ως προς συνθήκη της Λισαβόνας. Αν θέλουμε οι πολίτες να νιώσουν πιο, ότι βρίσκονται πιο κοντά, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τις ε, ε, αποφάσεις τους. Διαφορετικά στέλνουμε λάθος, αποστέλνουμε λάθος μήνυμα και δίνουμε λάθος στίγμα. Ο κύριος Βάτιμο. Ζητώ συγγνώμη και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο και βεβαίω συμφωνώ απόλυτα με όσα ανέφερε. Συμμετέχω, μάλλον με βρίσκει σύμφωνο η ανησυχία της πώς θα κατανοήσουν καλύτερα την Ευρώπη οι συμπατριώτες μας. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι στις τελευταίες ευρωεκλογέ είχαμε μία ε, πιο χαμηλή συμμετοχή των πολιτών. Και αυτό το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Βεβαίω όλα εξαρτώνται από τις αρμοδιότητες της Ευρώπης, διότι οι πολίτες αν, θα πρέπει να καταλάβουν αν αλλάζει κάτι στην καθημερινή του ζωή. Δηλαδή το πρόγραμμα Έρασμους έχει επιπτώσεις πολλοί γονείς στέλνουν τα παιδιά τους να σπουδάσουν αλλού και κατανοούν ότι κάτι αλλάζει. Επίσης με το ενιαίο νόμισμα, το οποίο δεν δέχτηκαν πολύ καλά όλοι. Στην Ιταλία διπλασιάστηκαν οι τιμές, άρα δεν ήταν θετικός ο αντίκτυπος. Το ζήτημα είναι ότι εάν υπάρχει αδυναμία δράσης από πλευρά, πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν γίνεται τίποτα. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Οι ψηφοφόροι μας ενδιαφέρονται για αυτά. Σε αυτά τα θέματα τι λέει η Ευρώπη. Η Ευρώπη σιωπά, γιατί δεν έχει αρμοδιότητες, δεν έχει εξουσίες. Χτες υπέβαλα μία επιστολή στην πρόεδρό μας εκφράζοντας την κατάσταση στην Ιταλία ως προς την ελευθερία τύπου. Βεβαίως ε, δεν ε, περιμένω η Ευρώπη να βομβαρδίσει την Ιταλία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει ένας αντίκτυπος. Όλα εξαρτώνται από τις εξουσίες της Ευρώπης και εμείς ως Επιτροπή Πολιτισμού ίσως κάτι μπορούμε να κάνουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο να προβάλλει κανείς πολιτική προπαγάνδα μέσω θεσμικών παρεμβάσεων. Δηλαδή, τι έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έπρεπε να αποκαταστήσουμε την τάξη. Είχαμε την ΕΚΑΧ. Κάτι άλλαζε. Και έπρεπε να ξεπεράσουμε το παρελθόν. Εμείς αν ε, προβαίνουμε σε μία πολιτική προπαγάνδα και λέμε «Α, η Ευρώπη είναι κάτι το καλύτερο, ο πολίτης θα πει «Μα τι αλλάζει την καθημερινή μου ζωή». Θα πρέπει η Ευρώπη να είναι πιο παρεμβατική σε θέματα που αφορούν τους πολίτες, μετανάστευση, κοινωνική αρρωγή, φορολογικές ελαφρύνσεις. Κάθε φορά που μιλάμε για την Ευρώπη μας λένε «Α, ναι, υπάρχουν όμως φορολογική παράδειση και τι θα γίνει». Σας το υπενθυμίζω διότι μου ήρθε στο νου όταν μιλούσατε εσείς, ε, κυρία Επίτροπε. Ευχαριστούμε τον κύριο Βάτιμο. Ο κύριος Σουίνι. Ευχαριστώ. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την ε, παρέμβασή σας, ε, διότι εκτιμώ την ε, δημοκρατική διαδικασία στη Σουηδία, την ε, γείτονα χώρα και υπήρξε μια εξαιρετική ε, πρακτική στη Σουηδία ως προς την καταψήφιση του ευρώ του 2003 στη Σουηδία. Αν και η πολιτική ελίτ έκανε ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ιδέα αρχικά. Άρα δεν, ε, δεν επιβάλλατε τη θέλησή σας του Σουηδούς. Αν δούμε όμως τι έγινε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ε, Ολλανδία, στη Γαλλία και στην Ιρλανδία είχαμε πολύ μικρές αλλαγές και τώρα η Ιρλανδία θα ψηφίσει ξανά για την ίδια τη συνθήκη. Δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας ως προς την συνθήκη. Αυτό δεν είναι μάθημα δημοκρατίας. Τα μαθήματά μα θα πρέπει να τα παίρνουμε από τη Σουηδία. Ε, δεν βλέπω το λόγο γιατί να ψηφίσει η Ιρλανδία μία δεύτερη φορά τη στιγμή που δεν έχει αλλάξει τίποτα επί τη ουσία. Εμείς τώρα έχουμε πληγεί από το ευρώ, ενώ η Σουηδία ευεργετήθηκε από την μη κύρωσή του. Μιλήσατε για την επικοινωνιακή πολιτική και για θέματα ηθαγένειας. Νομίζω ότι τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μαζί μας, θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία και μία ενεργό συμμετοχή και επικοινωνία με τους πολίτες. Στη Φιλανδία, ε, όταν οι άνθρωποι διαφωνούν, ε, υπάρχει ε, μία ε, πραγματική θετική θεώρηση από τους πολίτες. Εγώ έχω παρευρεθεί με άλλους ε, ευρωβουλευτές στην τηλεόραση όπου διαφωνούμε και αυτό προσελκύει περισσότερο τους πολίτες, ακόμα και αν υπάρχει δυσανεξία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Βάλστρομ για την εισήγησή της που ήταν απόλυτα σαφής ε, και καινοτόμος. Ορισμένοι συνάδελφοι έθιξαν τα ζητήματα που ήθελα να θίξω και εγώ. Βεβαίως αυτή η Επιτροπή θα είναι μεγάλη σύμμαχό σας για την προώθηση των γενικότερων στόχων, έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε μία επικοινωνιακή πολιτική που να βρίσκεται πολύ κοντά στους πολίτες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει και οι υπάλληλοι να επανέλθουν σε αυτό το κοινό σχολείο και έχει μεγαλύτερη σημασία από τα πολυμέσα κάτι τέτοιο. Υπάρχουν δύο πολιτικά ερωτήματα διότι η Ευρώπη θα πρέπει να επικοινωνεί διαφορετικά. Ο κύριος Βάτιμο μίλησε για ένα θέμα ουσίας που αφορά και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η Ευρώπη κινείται προς μια αύξηση εξουσιών που να έχουν μεγαλύτερη επίπτωση προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Εσύ είπατε κάτι το οποίο με βρίσκει σύμφωνο πώς ε, αντιστράφηκε το θέμα της ε, επικοινωνίας, δηλαδή ότι η επικοινωνία θα πρέπει να τάσεται υπέρ της ηθαγένειας, των καθηκόντων και των δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει ε, αυτός ο σύνδεσμος, να ενδυναμωθεί αυτός ο σύνδεσμος μεταξύ πολιτών και επικοινωνίας. Αυτό είναι το κυρίαρχο μήνυμα, διότι δεν έχει γίνει κατανοητό μέσα στα πλαίσια της επικοινωνιακής μας πολιτικής. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο πολίτης θα πρέπει να ξέρει τι σημαίνει για την καθημερινή του ζωή οι κοινέ αξίες. Το δεύτερο ουσιώδες ζήτημα είναι η Εξή δυνατότητα. Πολλές φορές η επικοινωνιακή πολιτική δεν είναι αποδοτική. Πολλές φορέ. λέμε ότι η Ευρώπη δεν αποτελεί νέο. Μιλάμε για το κόστος της μη Ευρώπης. Υπάρχει ο ευρωσκεπτικισμός, οι επιμέρους δυσχέρειες. Υπάρχει διαθεσιμότητα προς το διάλογο. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη αντίσταση. Αυτό το είδαμε στα δημοψηφίσματα, ακόμα και από χώρες που ευεργετήθηκαν από την Ευρώπη. Άρα δεν πρέπει να, κάνουμε, να πούμε τι κάνει η Ευρώπη, αλλά ποιο θα ήταν το κόστος της μη Ευρώπης. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα. Μιλήσατε για τις νέες γενναίες. Εμείς θα πρέπει να στοχοθετήσουμε τις νέες γενναίες και πιστεύω ότι ο προϋπολογισμός είναι ιδιαίτερα χαμηλός, όπως είπε η Επίτροπος, και ιδιαίτερα τα προγράμματα για τους Ευρωπαίους νέους. Τα προγράμματά μας για θέματα ευρωπαϊκής ηθαγένειας είναι πολύ περιορισμένα επίσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός έγινε διότι θα πρέπει να συμμεριζόμαστε την ε, πείρα μας με τους άλλους νέους της Ευρώπης στα πλαίσια των σχολείων και των νέων, καθώς και της τριτοβάθμιας. Μιλήσατε και ως προς τα δίκτυα, δηλαδή τη συμμετοχή των δικτύων οπτικοακουστικών, ραδιόφωνο, τηλεόραση και μιλήσαμε και για τα τοπικά δίκτυα, τα τοπικά ραδιόφωνα πώς προωθεί η Επιτροπή την συμμετοχή αυτών των δικτύων έτσι ώστε να μπορέσει κανείς να καρποθεί αυτή την επικοινωνιακή πολιτική σε περιφερειακό και εδαφικό ε, επίπεδο. Έχω ακόμα πέντε ομιλητέ, οπότε θα δώσω τώρα το λόγο στην ε, Επίτροπο, ώστε να μπορέσει να απαντήσει. Ε, σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να καλύψει όλα τα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Σα ε, ευχαριστώ όλου για τα σχόλιά σα και για τα ερωτήματα που μου θέσατε και θα προσπαθήσω να απαντήσω αυτά τα ερωτήματα σύντομα και ορθά. Καταρχήν, η κυρία Χέλγα Τρούπερ αναφέρθηκε στα management partnerships, ε, διαιτερικές ε, διαχείρισης ε, ως ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και πράγματι συμφωνούμε σε αυτό ότι θα πρέπει να κάνουμε για να δούμε δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε από κοινού στη Γερμανία, στη Σουηδία, ούτως ώστε να παράσχουμε καλύτερα τις πληροφορίες, να ακούσουμε καλύτερα τους πολίτες μας ε, και βέβαια μπορούμε να έχουμε πολύ διαφορετικές ε, προτεραιότητες. Σε κάποια κράτη-μέλη λένε ε, πω για παράδειγμα πρέπει να δώσουμε στου δασκάλου, στου εκπαιδευτικού τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παράσχουμε τέτοιε δυνατότητε εκπαίδευση, ενώ άλλα κράτη-μέλη εστιάζουν στη νεολαία, στους νέους μέσω άλλων, άλλου είδους δράσεων. Άρα λοιπόν αυτό το εργαλείο ήταν, αποδείχθηκε πολύ χρήσιμο. επιτρέψτε μου επίσης εδώ να υπογραμμίσω πως ένα τμήμα των δικό μου να αφορούσε και την, τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και όπως γνωρίζετε ε, εδώ και κάποιο καιρό αποστέλουμε όλες τις δικές μας προτάσεις στα Εθνικά Κοινοβούλια και είχαμε εκατοντάδες επισκέψεις από αντιπροσωπείες Εθνικών Κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα δεν έχουμε δει το αποτέλεσμα αυτή τη στενότερη συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια, αλλά είμαι πεπισμένο πω αυτό θα συμβεί. Δηλαδή θα το δούμε αυτό το αποτέλεσμα του να ενσωματώνεται μέσα στην καθημερινή συζήτηση ε, που γίνεται στα Εθνικά Κοινοβούλια Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνεται τελικά στην ίδια τη δημοκρατική κουλτούρα του κάθε κράτου μέλου. Ε, Ευρώπη. Ε, θεωρώ πως αυτό αποτελεί, θα αποτελέσει μεγάλη επιτυχία και, ό, και αν δούμε κάποια στιγμή την επικύρωση της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, τότε πράγματι θα έχουν πολύ σαφέστερο ρόλο τα εθνικά κοινοβούλια, θα έχουν ε, ένα πιο μεγάλο ρόλο να παίξουν ε, και θα πρέπει να είναι και ανάλογα προετοιμασμένα για να τον αναλάβουν. Οπότε υποστηρίζω τα όσα είπατε εν είδη αναγνώρισης όσο γίνονται σε, σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, Υπήρξαν τώρα αρκετοί ομιλητές που αναφέρθηκαν στα δίκτυα τα τηλεοπτικά και ραδιοφώνου, TV Radio Networks και ε, σας είπα πως γι' αυτό αποφασίσαμε ήδη και οριστικοποιήσαμε τη δική μας ε, ε, πολιτική στον χώρο Εικόνα και ήχο, audiovisual, γιατί ακριβώς δεν ε, αντιλαμβανόμαστε την Ευρώπη ως κάποιον ο θα πρέπει να παρέχει την ενημέρωση. Συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους δημοσιογράφους και αυτό που τους παρέχουμε είναι η ενημέρωση για να μπορούν να, ε, ε, αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή παρέχουμε τη μετάφραση και γενικότερα τους τρόπους τα όσα απαραίτητα για τη δημιουργία αυτών των δικτύων. Ήδη λοιπόν υπάρχει αυτό το δίκτυο σε σχέση με τα όσα μπορείτε να ακούσετε τόσο στο Βέλγιο αλλά και στις διάφορες χώρες σας έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ψηφιακών ειδήσεων, digital news όπου μπορείτε δηλαδή μέσω του διαδικτύου να αναζητήσετε τα πλέον ενδιαφέροντα άρθρα που καλύπτουν τις ευρωπαϊκές υποθέσεις επίσης εργαζόμαστε αυτή την περίοδο και ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ενός ε, δικτύου ομάδων ε, συγγνώμη, ε, τηλεόρασης ε, όπου προσπαθούμε να έχουμε τη συμμετοχή περίπου 200 τηλεοπτικών καναλιών για να παρέχουμε ακριβώς καλύτερες ειδήσει και ταυτόχρονα συνεχίζει βέβαια και το Europe by Satellite όπου παρέχεται α, χωρίς σχόλια απλώς και μόνο υλικό, τηλεοπτικό υλικό από το οποίο μπορούν να αντλούν ε, υλικό οι διάφοροι σταθμοί και έχουμε μάλιστα διπλασιάσει και τις δυνατότητες του Europe by Satellite ούτως ώστε ε, να έχουμε ε, να διαθέτουμε περισσότερο υλικό ταυτόχρονα όμως συνεχίζει να ισχύει και η συντακτική ουδετερότητά τους, η ανεξαρτησία τους. Ταυτόχρονα έχουμε το Euronews το οποίο ανήκει σε δημόσια τηλεοπτικά κανάλια ε, με ουδέτερο τρόπο και πάλι εδώ έχουμε προβλέψει συντακτική ανεξαρτησία ε, ε, το συμβόλαιο παροχή υπηρεσία με το Euronews θα λήξει σύντομα και θα γίνουν κάποιε συζητήσει στο πλαίσιο της ανανέωσης για να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Πάντως όλα αυτά συγκαταλέγονται στην πολιτική του πώ μπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και το διαδίκτυο, γιατί αυτά είναι τα τήρια κανάλια τη ενημέρωση το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν αποτέλεσαν σημαντικό τμήμα των δικών μα προσπαθειών τα τελευταία χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τον Ιρλανδικό λαό, ε, δεν τον σεβόμαστε. Φυσικά και όχι. Και προφανώ θα έχουν να, να, να, να πούνε κάτι, έχουν λόγο σε σχέση ε, με τη νέα συνθήκη τη Λισαβόνα. Αλλά γιατί πρότεινε η κυβέρνησή του να υπάρξει ένα νέο δημοψήφισμα. Γιατί αποτέλεσε αυτό το ζήτημα τόσο σημαντικό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θέλαμε να σεβαστούμε τα όσα μας είπαν. Θέλαμε να ακούσουμε το ποιος ήταν ο λόγος του, γιατί είπαν όχι στο δημοψήφισμά τους. Για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει κάποιος τρόπος για να διστεδάσουμε τις ανησυχίες ε, του ελληνικού λαού. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Δεν ήταν το ίδιο κείμενο της συνθήκες. Τα πιο, οι πιο σημαντικές ανησυχίες των Ελλάντων ελήφθησαν υπόψη και έτυχαν διαπραγμάτευσης με όλους τους άλλους ε, πολιτικούς ηγέτες και γι' αυτό είπαμε ακριβώς αφού επιλύσαμε το ζήτημα της άμυνας, των εκτρώσεων, όλα τα άλλα ζητήματα που απασχόλησαν τον ελληνικό λαό, θα ήσασταν σε αυτή την περίπτωση διατεθειμένοι να αποδεχτείτε. Γιατί σας υπενθυμίζω πως η εν λόγω συνθήκη έλαβε το ναι σε άλλα κράτη-μέλη. Άμα έχουμε λοιπόν 25 κράτη-μέλη στα οποία ήδη έχει λάβει η χώρα η πλήρη επικύρωση αυτή τη συνθήκη, δεν είναι σημαντικό να ληφθούν και εκείνοι υπόψη, να σεβαστούμε και τη δική του ε, στάση και να, να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν ε, τρόπο συνεργασία. Γιατί όπω γνωρίζετε, το σημείο αφετηρία για όλη αυτή τη συνθήκη ήταν να καταστεί η Ευρώπη πιο δημοκρατική, πιο αποτελεσματική και να έχει ε, να είναι πιο καλά εφοδιασμένη για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου. Όλοι οι κανόνες της συνθήκης Ε, είχε, ε, δηλαδή το όλο σκεπτικό είχε ξεκινήσει με, όπως οργανωνόταν μέχρι στιγμής στην Ευρώπη αφορούσε στο μισό αριθμό ε, κρατών μελών από ό,τι έχουμε σήμερα. Προφανώς λοιπόν ε, μα έχουν απασχολήσει όλε μα οι ανησυχίε ε, του Ιρλανδικού λαού και σε καμία περίπτωση δεν τον παρακάπτουμε και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να ε, διορθώσουμε τα σημεία εκείνα τα οποία προκαλούσαν ε, δυσκολίε στην Ιρλανδία. Αλλά θεωρώ πω είναι προ το συμφέρον ολόκληρη τη Ευρώπη να δημιουργήσουμε μια συνθήκη η οποία είναι απλούστερη, είναι δημοκρατικότερη, είναι αποτελεσματικότερη, ώστε να δούμε τελικά πώ μπορούμε να κάνουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε. Δηλαδή πώ θα αντιμετωπίσουμε την οικονομική κρίση, πώ θα αντιμετωπίσουμε τι κλιματικέ μεταβολέ, πώ θα διασφαλίσουμε την ενεργειακή ασφάλεια, των, δηλαδή των ενεργειακών μα ε, προμηθειών. Όλα αυτά τα ζητήματα θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε όντα πιο αποτελεσματικοί στον τομέα τη λήψη αποφάσεών μα. Ε, και θέλουμε και ε, ο ελληνικό λαό να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει και θα υπάρξει ένα δεύτερο ε, δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και προφανώς και θα τύχει σεβασμού και το ε, αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος. Ε, και νομίζω πως η κάθε κυβέρνηση θα έπρεπε να κάνει το ίδιο εφόσον έχει διοργανώσει ένα δημοψήφισμα, δηλαδή να σεβαστεί το αποτέλεσμα του. Τώρα, κύριε Βάτιμο, ε, ρωτήσατε, δεν έχει να πει κάτι η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία. Ε, ναι, ε, εμείς κάναμε πρόσφατα κάποιες δηλώσεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την ανάγκη ε, προστασίας ελεύθερου και ανεξάρτητου τύπου και μέσων ενημέρωσης και αυτό αποτελεί κύριο στοιχείο της δικής μας δουλειάς, δηλαδή διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία κοδομούν τη σημερινή Ευρώπη. Ε, υπάρχουν λοιπόν αρκετοί από εμά, επίτροποι, που προσπαθούν να παίξουν ένα ρόλο εδώ. Συμφωνώ μαζί σας ε, ως προς το ότι θα πρέπει να γίνει εδώ μια ζωντανή συζήτηση Δηλαδή αυτή η πολιτική σύγκρουση που υπάρχει, η διαμάχη, ε, είναι μέρος της πολιτικής συζήτησης και αν δείτε το δικό μου blog θα δείτε ότι ε, αφήνουμε εκεί να εκφράζονται ακόμα και πιο ακραίες απόψεις ε, και προτιμώ μάλιστα να, να πηγαίνω σε δημόσιες συζητήσεις για να δω, να συναντηθώ με αυτούς που λένε όχι, με αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη. Είναι σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα μιας πολύ πολύ ζωντανή συζήτηση. Αυτό αποτελεί παράδοση στι δικέ μα σκανδιναβικέ χώρε, αλλά νομίζω πω αποτελεί παράδοση και σε όλε τι υπόλοιπε. Ε, δηλαδή, δεν είναι ο σκοπό μα να κάνουμε του υπόλοιπου να σιωπήσουν, αλλά αντίθετα να του ε, ενθαρρύνουμε να συζητήσουν και να εκφραστούν τόσο τα υπέρ και τα κατά. Ε, τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Ε, μπορείτε να διαβάσετε όμως τις ε, μερινές ε, Ιταλικές εφημερίδες για να δείτε τι λένε εκεί και αν υπάρχει συζήτηση. Λέει ο κύριος Βάτιμα. Ναι, γνωρίζω πως πολύ συχνά οι δημοσιογράφοι λένε πως ε, είναι συνήθω βαρετά τα όσα συμβαίνουν στην Ευρώπη. Είναι δύσκολο να εξηγηθούν λόγω του περίπλοκου εδώ οικοδομήματο. Έχουμε να κάνουμε με τόσα ε, κράτη-μέλη όπου πρέπει να επιτευχθεί συνένεση. Άρα λοιπόν υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία που συνεγορούν κατά ε, το να συντάσσονται άρθρα και να γίνονται αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, ε, βέβαια, με τι απασχολούμαστε με νομοθεσία. Γενικά η νομοθεσία δεν δημιουργεί τόσο συναισθηματικέ αντιδράσει και ούτω καθεξή. Από την άλλη όμω πλευρά, τα όσα πράττουμε επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των απλών πολιτών στην Ευρώπη. Γι' αυτό και προσπαθούμε να μεταφράζουμε τα όσα εμεί αναφέρουμε ακριβώ σε συνέπειε ε, που θα υπάρξουν στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Γι' αυτό κάνω και τα έντυπά μα στα φυλάδια δηλαδή ω προ το πώ εγώ ω απλό πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νιώθω τον αντίκτυπο ή υφίσταμαι τι συνέπειε των όσων αποφασίζονται. Αποτελεί κάτι τέτοιο προπαγάνδα τίθεται το ερώτημα. Ε, εάν θέλει κάποιο ε, να χρησιμοποιήσει τον όρο προπαγάνδα, ουσιαστικά το κάνει και εκείνο χειριστικά. Δηλαδή προσπαθεί να φέρει εδώ αναμνήσει ε, ε τη Σοβιετική Ένωση ή, εν πάση περιπτώσει, να δημιουργήσει, να, να, δώσει μια αρνητική χρειά σε αυτό το έργο. Προπαγάνδα σημαίνει όμω ότι ελέγχει κανεί τα μέσα ενημέρωση και ελέγχει την παιδεία. Αλλά εμεί δεν κάνουμε κανένα από αυτά. Εμεί έχουμε ελεύθερο και ανεξάρτητο τύπο στην ε, Ευρώπη, ο οποίο έχει συνήθω επικριτική διάθεση απέναντί μας. Περισσότερες είναι επικρίσεις που δεχόμαστε από ότι τα αλληλούια, τα μπράβο δηλαδή ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε εσάς. Και σε καμία περίπτωση δεν ελέγχουμε καταστήματα παιδείας ε, στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη υπερασπίζονται ε, και πάρα πολύ μαχητικά τα δικά του συστήματα εκπαίδευση. Άρα λοιπόν συνήθω η κριτική που μα ασκείται είναι ότι είμαστε υπερβολικά βαρετοί. Γιατί παράγουμε νομοθεσία και προσπαθούμε να την εξηγήσουμε και φυσικά μερικέ φορέ είμαστε βαρετοί σε αυτό. Ε, αποτελεί κάτι τέτοιο προπαγάνδα, όχι. Όχι. Ε, γιατί ε, δεν θα γινόταν ανεκτή η προπαγάνδα. Οι άνθρωποι τη Ευρώπη δηλαδή δεν θα ανέχονταν να υπάρχει μια προπαγάνδα. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε τα πράγματα από την ε, ε, οπτική γωνία του πολίτη. Αποτελεί δικαίωμα του πολίτη να ενημερώνεται και να έχει λόγο σε όλα αυτά και να ασκήσει κριτική εφόσον το επιθυμεί. Αυτή τη δυνατότητα πρέπει να του παράσχουμε και αυτά είναι τα καλέ που του δίνουμε. Σας ευχαριστώ. Τώρα βλέπω ότι έχουμε 7 παρεμβάσεις. Σας παρακαλώ μην καταχραστείτε του χρόνου. Δύο λεπτά. Ο κύριος Μάρτιν. Καθώς, ε, κύριε Πρόεδρε, ε, περιορίσατε το χρόνο αγορευσής μας, θα, πω, θα περιοριστώ σε λίγα πράγματα μόνο. Ε, ως ε, άνθρωπος ο οποίος τάσεται κατηγορηματικά υπέρ της Ευρώπης ε, σας θεωρούσα πάντα ως έναν από τους κύριους αντιπάλους μας ε, και αυτό δεν είναι προσωπικό απέναντί σας. Ε, πάντα εκτιμούσα τι δικέ σας, ε, τις δικές σας προσπάθειες. Ε, και δεν αποτελεί σήμερα το γεγονός ότι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι αποτελώ πλέον μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού. Και αυτό γιατί θεωρώ πως πολλά σημαντικά πράγματα δεν επιλύθηκαν. Από αυτό δηλαδή που διαπιστώνουμε σε δημοσκοπήσεις ε, σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό πνεύμα, την, ευρωπαϊκή ιδέα ε, και τα όσα διαπιστώνονται εκεί ίσως προβλήματα. Αφενός. Και μετά μα δούμε και τα όσα ε, συμβαίνουν ε, σε σχέση με τον εξοραϊσμό και με τις προσπάθειες να μην ε, ακούγονται κριτικές απόψεις, τότε θα διαπιστώσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια γενικότερα διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων και δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο G2 Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα αλλά G3 Ηνωμένε Πολιτείε και Κίνα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, πρέπει να γίνει κάτι εδώ και βλέπω ότι έχετε μια καλή αρχική προσέγγιση, αλλά, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Μας είπατε ότι σε ό,τι αφορά ε, την, γενικά τις χώρες της Ευρώπης έχει γίνει ε, μια είχε γίνει μια ε, πολύ μεγάλη συζήτηση ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα εμεί στη δική μου χώρα έγινε τόσο μεγάλη συζήτηση που καταφέραμε να αυξήσουμε την προσέλευση τη κράτου κατά 6%. Όμως εκείνο που δεν ισχύει είναι ότι ε, πράγματι προωθήθηκαν οι ζωντανές συζητήσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα όπου υπάρχουν ευρωπαϊκές υπηρεσίες οι οποίες προσπαθούν να, να αποτρέψουν το να λαμβάνουν χώρα τέτοιου είδους ζωντανές συζητήσεις υπάρχουν περιπτώσεις όπου άτομα τα οποία ε, προσπαθούν να ασκήσουν κριτική ε, γίνονται προσπάθειες να αποσιωπηθούν ακόμα και ε, και στο ίδιο αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και άλλοι οι οποίοι απλά προσπαθούν να κάνουν επικοδομητική κριτική. Ε, ε, μετά υπήρχαν κάποιε καταγγελίε ότι προσπαθεί, ε, καταβάλει μάλιστα χρήματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ώστε να γίνουν έτσι αποσυμπήσει ή χρηματοδοτεί την εκπώνηση άλλων τοποθετήσεων. Και έχω πάρα πολλές εκθέσεις εδώ να σας δείχνω πόσο ε, πραγματικά πολύ μεγάλες πιέσεις άσκησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ώστε ε, να καταρτίζονται ε, θετικές εκθέσεις και αυτό καταδεικνύει ότι δεν ακούσατε τα όσα θέλαμε να σα πούμε. Ε, και ελπίζω ο ή η διάδοχό σα ε, θα, προσπαθήσει να κάνει περισσότερα πράγματα και δεν απευθύνομαι σε εσά προσωπικά. Γνωρίζω πόσα προσπαθήσατε να κάνετε. Αλλά σα λέω ότι ασκήθηκαν πάρα πολύ μεγάλε πιέσει, πράγμα που με τη σειρά του βέβαια δημιουργεί μια πάρα πολύ επικίνδυνη πόλωση. Γιατί λέει κανεί ότι είσαι μαζί μας ή είσαι εχθρός μας, είσαι αντίπαλός μας, είσαι κατά των όσων προσπαθούμε να κάνουμε. Και κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, και το οποίο δηλαδή ε, ε, ε, υπάρχει ανάγκη για να γίνει εδώ μια μεγάλη μεταρρύθμιση, σε... αφορά το διαδίκτυο. Δηλαδή ενημέρωση, γιατί ο πολίτη θέλει να μάθει πού μπορώ να συμμετάσχω, σε τι, πώ μπορώ να λάβω την τάδε επιδότηση, τι χρειάζεται να κάνω. Εκεί δεν υπάρχει το υλικό, θα πρέπει να γίνουν πολλά σε αυτό το τομέα ε, και νομίζω πως αυτός τουλάχιστον είναι ένας στόχος ο οποίος είναι κοινός και για μένα και για σας. Πρόεδρος είναι εκτός ε, μικροφώνου δυστυχώς. Ήθελα να πω πως υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι πληρώνονται για να ασκούν προπαγάνδα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι υπέρ αυτής. Ο κύριος Λόκογκαρτ, αντιπρόεδρος παρακαλώ. Oh, jeg er medlem, og det, er det vil sige, at Jeg hører den fra Venstrøm, og jeg er- Άκουσα, άκουσα κυρία Βάλστρομ, είμαι πάρα πολύ εντυπωσιασμένος για τη δέσμευση της θέσης και τα αποτελέσματα τα οποία επιτύχατε. Νομίζω ότι όντως είναι το αποτέλεσμα μιας σκανδιναβικής παράδοσης που γνωρίζω και της οποίας αποτελώ μέρος ως πρώην δημοσιογράφος. Δεν θα ήθελα να κάνω μια μεγάλη πολιτική δήλωση σχετικά με τη θέση μου για αυτή την κατάσταση, αλλά υπάρχουν ε, ορισμένα ε, συγκεκριμένα θέματα τα οποία θα ήθελα να θέσω. Έχω μια κάποια πείρα σχετικά με τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν έρευνες σχετικά με τις πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν και ποιες ήταν οι επιπτώσεις τους. Όταν προσπαθούμε να δούμε ποια ήταν τα αποτελέσματα, έχουμε πληροφορίες, έχουμε στοιχεία και νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που ακούω εδώ που βασίζονται σε προσεγγίσεις, μεθόδους, πολιτικές υποκασίες. Χρειαζόμαστε τις απαιτούμενες γνώσεις που να δείχνουν ποια είναι η πραγματική κατάσταση και ποια είναι τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν πραγματική επίδραση πάνω στον πληθυσμό. Πιστεύω επίσης ότι ο ευρωπαϊκός χώρος είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να λάβουμε ε, πρωτοβουλίες, υπάρχουν όλα τα τεχνολογικά μέσα, το διαδίκτυο, ε, τα κανάλια τηλεόρασης, ραδιόφωνο, αλλά θα πρέπει να έχουμε κάτι το ευρωπαϊκό. Δεν πρόκειται απλώς για μια δράση σε επίπεδο πολιτικό. Θα πρέπει να παρεμβαίνει και η κοινή γνώμη. Πώς η Κομισιό θα κατορθώσει να έχει μια ευρωπαϊκή κοινή γνώμη έχουν αναλυθεί πρωτοβουλίες για να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Μιλάμε συχνά για ε, να προκληθεί ένα κοινό ενδιαφέρον. Θα έπρεπε ίσως να έχουμε ορισμένα δημοψηφίσματα κοινά, ψηφοφορίες κοινέ, εκλογές κοινέ. Θα έπρεπε ίσως να ψηφίζουμε μαζί για έναν επίτροπο, για έναν πρόεδρο για να δημιουργήσουμε ορισμένες πρωτοβουλίες, ορισμένες δράσεις, ούτω ώστε οι άνθρωποι που θέλουν να δεσμευτούν να μπορούν να το πράξουν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Επίτροπε, συγγνώμη, ε, για, τις, τα όσα μας παρουσιάσατε σήμερα εδώ. Σας άκουσα με μεγάλη προσοχή και Ε, άκουσα να την ανησυχία πως ε, δεν λαμβάνουμε επαρκώς υπόψη μας τους ε, πολίτες μας. Όμως εγώ θεωρώ πως ιστορικά, διαχρονικά η ευρωπαϊκή αίσθηση των πολιτών μας αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο. Όμως, εάν κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης, μεταξύ νέων δηλαδή, και παλαιών κατομελών, ε, θα δούμε πως υπήρξαν μεγάλες διαφοροποιήσεις, διαφορές σε ό,τι αφορά την προσέλευση στις κάλπες. Εγώ προέρχομαι από τη Σλοβενία, ε, αλλά ε, διαπίστωσα ότι και σε άλλα νέα κράτη-μέλη η προσέλευση ήταν πολύ χαμηλή. Η συμμετοχή δηλαδή στις ευρωπαϊκές εκλογές. Εμεί είχαμε και την και ε, πρόσφατα και την ε, Προεδρία του Συμβουλίου και παρόλα αυτά η κατάσταση δεν άλλαξε. Δηλαδή η προσέλευση κάλπες παρέμεινε πολύ χαμηλή. Έχετε προβλέψει κάποια ιδιαίτερη στρατηγική για αυτές τις χώρες στις οποίες δηλαδή αυτή η διάσταση ε, είναι πιο προβληματική. Δηλαδή δεν έχει ακόμα επέλθει στον πληθυσμό αυτή η ταύτιση με την Ευρώπη. Μήπως θα μπορούσαμε για παράδειγμα να επέμβουμε στην παιδεία, στα όσα διδάσκονται, στην ύλη δηλαδή τη διδασκόμενη. Ε, Προφανώς δεν μπορούμε να παρέμβουμε εδώ σε ζητήματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία των κρατομελών, αλλά μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη σε προσπάθειες που θέλουν να κάνουν. Ε, και νομίζω πως αυτό αποτελεί ε, καθήκον μας. Θεωρώ πως θα μπορούσαμε με έναν ήπιο τρόπο να πείσουμε τους πολίτες μας πως η ταύτισή τους με την, με την Ευρώπη δεν έρχεται σε αντίθεση με την ε, ταυτότητά τους ως πολίτες της δικής τους χώρας. Μπορώ δηλαδή να είμαι πολίτης τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χώρας μου. Δεν είναι αλληλοαποκλειόμενα σε αυτές οι δύο ιδιότητες. Αλλά πώς μπορούμε να τους το καταστήσουμε αυτό σαφές. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για όλους μας, αποτελεί ζητούμενο. αλλά θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι έχει και πολιτική, ε, πολιτισμική συγνώμη, διάσταση η Ευρώπη. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα, ε, ένας ε, πόλος εξουσίας και πολιτικής. Ευχαριστούμε κυρία ε, Επίτροπε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο πτυχές. Ε, είπατε πως, πως νέα ε, στρατηγική επικοινωνίας ε, ε, έχει περιλάβει και την δημιουργία νέων τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών ειδικότερα εφόσον καλύπτονται πτυχές οι οποίες είναι πολύ σημαντικές για τους πολίτες. Εδώ το ζητούμενο είναι η επικοινωνία, δηλαδή προσπαθούμε δηλαδή να καταστήσουμε τα πάντα πιο κατανοητά για τον πολίτη. Άρα λοιπόν αυτό που θα ήθελα να σας καλέσω είναι ε, να κάνετε είναι να συμμετάσχουν σε αυτά τα νέα δίκτυα, τα τηλεοπτικά, τη ραδιοφωνικά δίκτυα και οι ε, ε περιφερειακοί και τοπικοί ε, οργανισμοί τοπική αυτοδιοίκηση δηλαδή, γιατί πραγματικά έχουν να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, την ποιότητα και τελικά τη σαφήνεια του μηνύματο που προσπαθούμε να περάσουμε. Αναφερθήκατε εδώ ε, σε μια ε, ορισμένη διάσταση ως προς το πώς ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το διαδίκτυο και να το αξιοποιήσουμε ως ένα εργαλείο για να μας βοηθήσει στη μεγαλύτερη προσέλευση στις κάλπες. Εδώ βέβαια προφανώς η κάθε χώρα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά έχει το δικό της τρόπο οργάνωσης, αλλά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές Και αφού βρισκόμαστε σε, σε φάση ακριβώς ε, εφαρμογή τη συνθήκη της Λισαβόνα, θα πρέπει να διασφαλιστεί το δικαίωμα για όλου του πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφίσουν μέσω του διαδικτύου σε αυτές τις επόμενες ε, κοινοβουλευτικέ εκλογέ. Ε, και επίσης θα ήθελα να τονίσω πως ε, ε, μία από τις ε, λιγιακές ομάδες στις οποίες είναι πάρα πολύ χαμηλή η συμμετοχή στη πληροφορία στις εκλογές είναι αυτή κάτω των 25 ετών. Οπότε ίσως θα μπορούσαμε να εστιάσουμε λίγο και τις λύσεις που προσπαθούμε να βρούμε στα κράτη-μέλη εκεί. ο δικός μας πρόεδρος ε, άσκησε το δικαίωμα αρνησικηρίας του κατά της εξέβρεσης μιας τέτοιας λύσης παρότι η κυβέρνηση είχε ταχθεί υπέρ, αλλά θεωρώ πως πραγματικά μία τέτοια δυνατότητα, δηλαδή μέσω του διαδικτύου, ε, θα, μπορούσε, θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τι επόμενε ευρωεκλογέ ε, για όλους τους πολίτες, οπότε θα ήθελα να σας καλέσω να το ε, επιτύχετε αυτό. Thank you, uh, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε θα ήθελα να σας συγχαρώ για τα όσα ε, μας είπατε και για τον ενθουσιασμό σας που από τη δική μου την προοπτική, από ε, την δική μου την πλευρά δεν είναι από τα ευκολότερα έργα. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ήταν οι ευρωεκλογές, τις οποίες όλοι ζήσαμε και είπαν, λέχθηκαν τόσα πολλά πράγματα από άλλους ε, της Επιτροπής και δεν μίλησαν πάντοτε για ευχάριστες εμπειρίες. Το θέμα που αναφέρθηκε από πολλούς είναι ένα θέμα κλειδί. Εμείς ως ευρωβουλευτές είμαστε υποτίθεται μια, ένας δημοκρατικός ε, θεσμός. Αλλά όταν ε, δεν υπάρχει μεγάλη συμμετοχή στις εκλογές, αυτό ε, νομίζω μειώνει την δημοκρατική μας αξιοπιστία. Είναι ένα θέμα κλειδί λοιπόν για όλους μας. Και με ενδιέφεραν οι 11 χώρες όπου η συμμετοχή αυξήθηκε. Ποιες είναι αυτές οι χώρες, θα με ενδιαφέρε να μάθω. Και επίσης το σχόλιο σας ότι όταν γίνεται προεκλογική εκστρατεία για θέματα ευρωπαϊκά, αυτό αυξάνει τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα περισσότερα για το θέμα αυτό, γιατί αυτό ε, είναι αντίθετο με τα όσα ακούμε πολλές φορές, ότι δεν είναι, οι άνθρωποι δεν ψηφίζουν για τα ευρωπαϊκά θέματα και δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτά. Ε, μας ενδιαφέρει για το τι ψηφίζουν. Ίσως να μας πείτε μερικά πράγματα. Κάποιος από τους προηγούμενους ομιλητές μίλησε για την ηλεκτρονική συμπεριφορά. Θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερα για το θέμα αυτό, γιατί αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Χάκολα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ Ευχαριστώ την Επίτροπο Βάλστρομ. Άκουσα με πάρα πολύ προσοχή, παρακολούθησα με πάρα πολύ προσοχή τα όσα κάνατε τα τελευταία χρόνια ως Επίτροπος. Και εάν επιτύχετε μια δεύτερη εντολή θα είναι πάρα πολύ καλό. Ιδαλλιώ σας ευχαριστώ για την δουλειά που κάνατε μέχρι τώρα. Εξετίμησα ιδιαίτερα το γεγονός ότι Αναφερθήκατε στον σεβασμό της διαφορετικότητας, της ποικιλομορφία, ότι πρέπει να έχουμε συζητήσεις. Δεν υπάρχει ε, καμία άποψη σωστή, λανθασμένη για την ευρωπαϊκή πορεία. Απλώς υπάρχουν απόψεις διαφορετικές. Με τον ένα ή άλλο τρόπο, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν μας αρέσουν ε, τα μπλοκ που μας φέρνουν την αντίφαση, τα περιθωριοποιούμε. Αυτή είναι μια κακή βάση ανάπτυξης για τη συζήτηση. Μας λένε ότι εμείς είμαστε Ευρωπαίοι πρεσβευτές, αλλά πρέπει να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε, πώς μεταχειριζόμαστε των πλησίων μας, πώς μεταδίδουμε αυτήν την εικόνα στους ψηφοφόρους, στους πολίτες και μέσα στο Κοινοβούλιο υπάρχει ένα χάσμα, ένα χάσμα ανάμεσα στους διάφορους βουλευτές και αυτό αντανακλάται νομίζω και στα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε οι ψηφοφόροι να κουνηθούν, να πάνε, να ψηφίζουν. Χρειάζεται λοιπόν μια πραγματική ε, συζήτηση επικοιλόμορφη που να συμπεριλαμβάνει και την αντίφαση. Για να κλείσω με αυτές τις ευχαριστίες θα έλεγα ότι απαντήσατε καλά στα όσα λέχθηκαν και σε αυτά που σας ζητήθηκαν για την Ιρλανδία μου θυμίζει το τραγούδι του Elvis Costello ότι ήταν σαν μια συνάντηση στην ενορία όπου όλοι ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι αλλά αυτό που θα έπρεπε και αυτό που πρέπει να κάνουμε για τη Σουηδία για όλους για να γνωρίσουμε, για να ε, πείσουμε τους Σουηδούς να μπουν στο ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό για μας τους Φιλανδούς, θα το καταλάβετε ε, κυρία Επίτροπε, τι μπορεί ε, να κάνει η Ευρώπη ούτως ώστε η Σουηδία να υιοθετήσει το ευρώ. Δύο ακόμα μιλητές έχουμε. Ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, καταρχήν σα ευχαριστώ για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πολυεπίπεδη παρουσίαση, η οποία κατέδειξε πόσε δυνατότητε πρωτοβουλία ε, έχουν ήδη ε, ληφθεί στο παρελθόν, ώστε να προσπαθήσουμε να ε, φέρουμε λίγο πιο κοντά την Ευρώπη στου πολίτε μα, να του ενημερώσουμε όσο στη δουλειά που γίνεται και ποια πλεονεκτήματα τελικά υπάρχουν για αυτού. Εγώ προέρχομαι από μια ε, προέρχομαι από μια περιοχή η οποία βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τα Βέλγιο και τις ε, κάτω χώρες και βλέπουμε εκεί πάντα να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ε, διάσταση και ακούω στον τελευταίο καιρό πως πράγματι αναγνωρίζουν οι άνθρωποι τα πόσα καλά έχει κάνει για αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η αίσθηση του ότι πράγματι ανήκουν στην Ευρώπη δεν υπάρχει δηλαδή για αυτούς η Ευρώπη είναι γραφειοκρατία, είναι διατάξεις, είναι κάτι το αρνητικό και αυτή η εικόνα τους δίνεται ξανά και ξανά μέσα των μέσων ενημέρωση και ίσω και από εμά του ίδιου, γιατί δεν ε, δίνουμε ακριβώ, δεν περνάμε αρκετά μηνύματα διαφορετικά από αυτό. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν πώ μπορούμε να επέμβουμε σε αυτή την εικόνα η οποία περνιέται ξανά και ξανά από τα μέσα ενημέρωση όπου παρουσιαζόμαστε δηλαδή ω γραφειοκράτε οι οποίοι απλά παράγουν διατάξει. Ε, και όχι απλά να, να υπερβούμε αυτή την εικόνα, αλλά να δούμε τι ακριβώς λείπει τελικά από τους πολίτες. Ε, πολλές φορές δηλαδή βλέπουμε δεν υπάρχει ενημέρωση και τελικά μένει μόνο η κριτική. Αυτή γίνεται αντιληπτή τουλάχιστον μόνο από τους ε, πολίτες ε, ε, χωρίς να, να, να γίνονται αντιληπτά τα θετικά τα οποία απλά θεωρούνται αυτονόητα τα οποία τα βιώνουν μέσα στην καθημερινότητά τους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξουν περισσότεροι πολλαπλασιαστές εντός εισαγωγικών οι οποίοι θα τονίσουν περισσότερο τα θετικά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εκεί υπάρχει πραγματικά ένα κενό μέχρι στιγμής. Κύριε Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ για τον τρόπο που προεδρεύσατε μέχρι τώρα τη συνεδρίαση και ευχαριστώ επίσης την κυρία Επίτροπο για την παρουσίαση της σήμερα το πρωί. Πάρα πολλά λέχθηκαν για την Ιρλανδία, έρχομαι από την Ιρλανδία, λέχθηκαν πολλά και για τη συνθήκη της Λισαβόνας η άρνηση της συνθήκης την τελευταία φορά στο δημοψήφισμα είναι κλασικό παράδειγμα έλλειψης επικοινωνίας, διότι όπως επεσήμανε και η κυρία Επίτροπος, οι εγγύησεις που δόθηκαν, ε, δόθηκαν ε, για κάτι που δεν ήταν στη συνθήκη ε, για, την, για τις για την απόξεση, για την, στο στρατιωτικό θέμα και γι' αυτό ψηφίσαμε όχι. τώρα υπάρχει κάποια διόρθωση, διορθώθηκαν τα πράγματα και στις 2 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε μάλλον ναι. Αν ψηφίσουμε ναι, σημαντική αλλαγή στη συνθήκη είναι ότι δίνει αρμοδιότητα για τον αθλητισμό και θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη τα οποία ψήφισαν μια αύξηση των πόρων για τον αθλητισμό. Η ερώτηση για την Επίτροπο. Εάν έχουμε αρμοδιότητα για τον αθλητισμό, ε, πώς θα αυξήσουμε την επικοινωνία ούτε ώστε να πλησιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους λαούς. Υπάρχει μια στρατηγική για την ε, προώθηση της συμμετοχής στον αθλητισμό, στα, στα σπορ, διότι εκεί νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ως μέλος της Επιτροπής θα ήθελα να πω δύο λόγια. Κάποιος είπε πως θα ήταν σημαντικό να δείξουμε κάπως στους ε, πολίτες μας ε, το τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ίσως θα μπορούσαμε να τους ε, ευαισθητοποιήσει με καλύτερο τρόπο. Κύριε Κώστα, νομίζω το είπατε. Νομίζω το είδα αυτό κάπου να γίνεται στην προεκλογική εκστρατεία. Και θα ήθελα να σας το προτείνω να το κάνετε. Αφήστε τους ανθρώπους να σκεφτούν τι θα συνέβαινε εάν δεν υπήρχε η Ευρώπη και να προβάλλεται αυτό μέσα το, στη τηλεόραση. Με κάποια παραδείγματα. Για να δώσουμε ένα ερέτημα στη σκέψη του πολίτη. Γιατί δεν το κάνει αυτό ποτέ. Γιατί κατά κάποιο τρόπο εμείς όσοι κατοικούμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε θύματα της επιτυχίας μας. Ό,τι έχουμε επιτύχει, το έχουμε επιτύχει και δεν το σκεφτόμαστε περαιτέρω, όπως είπε και η κυρία Χάνη. Δεν βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι, πόσο θετικό είναι. Δεν μας φαίνεται α, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Αυτή ήταν η δική μου πρόταση προς εσάς και σας δίνω το λόγο κύριε Βάζστρομ για να απαντήσετε στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχαριστίες και για την αναγνώρισή σας και για τις ε, ουσιώδεις ερωτήσεις που υποβάλατε. Και θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα από αυτά τα βασικά ζητήματα. Πώς ε, δημιουργεί κανείς μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα, σφαίρα επιρροής ίσως. Υπάρχουν τρία στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα διότι η λήψη αποφάσεων έχει προωθηθεί. Λαμβάνουμε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη συνέχεια πρέπει να έρθουμε σε επαφή, να φέρουμε σε επαφή αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις με τους πολίτες. Χρειάζεται μία πολυπολιτισμική ταυτότητα. Θα πρέπει δηλαδή να ενσωματώσουμε όλα αυτά τα ζητήματα στις καθημερινές μας συζητήσεις. Δηλαδή να έχουμε ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης. Αυτό θα πρέπει να είναι μια φυσική συνιστόσα της πολιτικής συζήτησης. Χρειάζεται μια, ένας πολιτισμός πολυμέσων. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε μια συζήτηση για τη νέα συνθήκη στην Ιταλία, Φιλανδία ή Σλοβενία. Πού και πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Τη στιγμή που δεν εντάσσεται στα καθημερινά μας νέα, μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτή την, αυτό το πολιτισμό πολυμέσων θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους δημοσιογράφους να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολλές φορές παραπονούνται ότι δεν κατανοούν τι συμβαίνει εδώ. Έχουμε ένα κέντρο τύπου όπου προβάλλουμε και κατάρτιση για επαγγελματίες δημοσιογράφους. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ε, αυτονομία τους, έτσι ώστε να μην προβούν, να μην έχουν δογματικές θέσεις. Υπάρχει λοιπόν αυτή η κατάρτιση, αλλά θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μέσω αυτών των δικτύων μπορούμε να δράσουμε και στο διαδίκτυο ή αλλού για να προβάλλουμε την ε, ευρωπαϊκή συζήτηση στα ΜΜΕ. Επίσης, πού συναντώνται οι πολίτες τα γραφεία ε, αντιπροσωπείας μας πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Είναι ευρωπαϊκή οίκη όπου προσπαθούμε να ανοίξουμε αυτούς τους ε, ε, οίκους έτσι ώστε να μην αποθηκεύουμε φύλαδια, αλλά να υπάρχουν εκθέσεις για την Ευρώπη, να οργανωθούν συναυλίες, να υπάρχει μια μικρή βιβλιοθήκη ή μια ζωντανή συζήτηση για ευρωπαϊκά θέματα. Έχουμε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες και θέλω να τονίσω ότι έχουμε αλλάξει με αυτή τη διαδικασία αποκέντρωσης. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε τα πάντα από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να κινηθούμε σε τοπικό επίπεδο. Και υπάρχουν αυτά τα κέντρα συνάντησης. Πρέπει να συνεχίσουμε ε, θα ήθελα να πω στον κύριο Μάρτιν ότι δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο. Έχουμε να κάνουμε με 27 κράτη-μέλη. Με όλα τα θεσμικά, με όλα τα γραφεία γίνονται πολλά σφάλματα και έχουμε παραδείγματα κακής ε, πρακτικής. Πρόκειται για μια αμφίδρομη πορεία. Πολλές φορές υπάρχουν ε, οι επικριτές που υπερβαίνουν κάθε όριο. Βεβαίως ε, διαπράττονται σφάλματα, δεν είμαστε τέλειοι, αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση πρέπει να είναι η σωστή και ο πολίτης έχει δικαίωμα να γνωρίζει, να πληροφορείται, να έχει μία φωνή. Γι' αυτό μιλώ για δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν αρέσουν σε όλους. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη ή μέλη, κυβερνητικά μέλη που θεωρούν ότι πρόκειται για μια πρακτική υπέρ των κυβερνήσεων και θα πρέπει να σιωπούν τα θεσμικά όργανα, να μην έχουν άμεση επαφή με τους πολίτες. Αυτό είναι αντιδεοντολογικό και παλιωμοδίτικο αν θέλετε. Οι πολίτες θέλουν να διαβουλεύονται ως προς τις βασικές μας προτάσεις, θέλουν να έχουν λόγο και μπορούν να το κάνουν διότι έχουν πληροφόρηση μέσω διαδικτύου. Έχουμε υπερβεί την ιδέα όπου έχουμε εθνικούς δήμους, έχουμε έναν ευρωπαϊκό δήμο και τα ΜΜΕ είναι διασυνοριακά όλο ένα και περισσότερο. Αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε και εσείς διαδραματίζετε σημαντικό ρόλο ως μέλη αυτής της Επιτροπής. Εσείς θα είσαστε στην εμπροστοφυλακή. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτά τα τρία στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα. Κάποιος πρέπει να είναι υπέρμαχος, συνεχής υπέρμαχος αυτής της γραμμής. Και βεβαίως μέσω των γραφείων ε, αντιπροσωπιών, αντιπρο, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να έχουμε σε επαφή με τα τοπικά μέσα, τους τοπικούς φορείς. Εάν μεταβείτε σε ένα κράτος μέλος, οι συνάδελφοι μεταβαίνουν καταρχήν στην πρωτεύουσα. Αλλά αν πάτε στο Κόρκ και μην, δεν παραμείνετε στο Δουβλίνο, θα έχετε καλύτερη κάλυψη από τον τοπικό τύπο θα συναντηθείτε με άλλους επιτόπιους φορείς. Προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε τα περιφερειακά και τοπικά μέσα πιο αποτελεσματικά. Άκουσα αυτά που είπατε σε σχέση με τα εκλογικά αποτελέσματα. Ίσως εσείς και η κυρία Πακ θα μπορούσατε να αναλάβετε μια πρωτοβουλία σε αυτή την Επιτροπή να οργανώσουμε ένα σεμινάριο όπου να εξετάσουμε τα αποτελέσματα των εκλογών. Έτσι ώστε εμπειρικά να δούμε τι συμβαίνει με το ευρωβαρόμετρο, να έχουμε όλα τα στατιστικά στοιχεία, έτσι ώστε να διοργανωθεί μία συζήτηση, ουσιώδη συζήτηση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών Συμμερίζομαι την απόψή σας ότι θα πρέπει να υπάρχει και το e-voting, η τηλεψηφοφορία. Διότι σε πολλά κράτη-μέλη δεν μπορούμε να ψηφίσουμε δια του ταχυδρομείου. Στη Σουηδία και στην Εσθονία υπάρχει το, η τηλεψηφοφορία, το e-voting και στη Σουηδία υπήρχαν και ε, υπενθυμίσεις ότι μπορεί κανείς να ψηφίσει σε αυτά τα κινητά λεωφορεία. Μπορούμε να πλουστεύσουμε τα πράγματα. Έχουμε ένα πεπαλαιωμένο σύστημα σήμερα το οποίο πρέπει να εξυγχρονίσουν τα κράτη-μέλη. Αλλά όλα εξαρτώνται από την εθνική πολιτική συζήτηση. Τα πολιτικά κόμματα και ομάδες φέρουν την ευθύνη. Αυτά που θα κάνουν θα προσδιορίσουν την υψηλή χαμηλή αποχή. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες ως προς τη διευκόλυνση της ψηφοφορίας, ιδιαίτερα για τους νέους. Άρα πολλοί είπαν ότι αν υπήρχε η τηλεψηφοφορία, το e-voting θα είχαν ψηφίσει. Προσπαθήσαμε μέσω MTV και άλλων καναλιών να, να επικοινωνήσουμε με τους νέους, να τους υπενθυμίσουμε για τις ημερομηνίες ε, ψηφοφορίας, για τη διεξαγωγή, αλλά δεν αρκεί αυτό. Δεν πρέπει να φαίνεται ότι προωθούμε κυβερνητικά ζητήματα, ή κατά της κυβέρνησης θα πρέπει να έχουμε μία ευρωπαϊκή συνιστόσα. Αλλά τα κόμματα που είχαν μία ευρωπαϊκή ατζέντα και εκεί όπου τα μέσα βοήθησαν σε αυτό είχαμε χαμηλότερη αποχή, μεγαλύτερη συμμετοχή. Θα πρέπει να προβούμε σε μία εις ανάλυση για να δούμε ποιοι ήταν οι βαθύτεροι λόγοι αποχής. Δεν ξέρω κατά πόσο ξέχασα κάτι. Ίσως οι Φιλανδοί μπορούν να πείσουν τους Σουηδούς να προσχωρήσουν στο ευρώ. Εγώ ήμουν δραστήρια στην εκστρατεία αυτή. Όχι ότι βοήθησε. Και όλα τα πολιτικά κόμματα υποσχέθηκαν να τηρήσουν, να λάβουν υπόψη την έκβαση του δημοψηφίσματος μακροχρόνια. Και αυτό το τηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δείτε την Ιρλανδία, Γαλλία και Ολλανδία, όταν ρωτήσαμε τους πολίτες και τους ρώτησαμε γιατί ψήφισαν υπέρ ή βλέπουμε ορισμένα κοινά στοιχεία. Πολλοί λένε ότι δεν θεωρούν ότι είχαν επαρκείς πληροφορίες. Δεν κατανόησαν επαρκώς τα επιμέρους ζητήματα, δηλαδή ε, δεν μπορούν να διαβάσουν όλα τα νομοθετικά κείμενα, τα ογκώδη κείμενα. Επίσης υπάρχουν εθνικά στοιχεία τα οποία επηρέασαν, αλλά και συγκεκριμένες ανησυχίες όπως στην Ιρλανδία. Και Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Θα πρέπει να τα σεβαστούμε όλα αυτά και λέμε. Ας δούμε αν μπορούμε να διορθώσουμε αυτά τα κακό κείμενα έτσι ώστε να έχουμε κάτι το οποίο θα επηρεάσει την υπόλοιπη Ευρώπη. Γι' αυτό προσβλέπουμε στην Ιρλανδία να μας βοηθήσει ήταν μια μακροχρόνια διαδικασία που αφορούσε όλα τα κράτη-μέλη. Είχαμε δύο δημοψηφίσματα όπου αποφάνθηκαν θετικά στη συνταγματική συνθήκη. Θα το σεβαστούμε αυτό. Τι θα κάνουμε με αυτούς που υπερψήφισαν. Οι επικεφαλής κρατών θα πρέπει να ακούν οι μεν τους δε. Δεν ξέρω αν έχουμε ένα σχέδιο για τον αθλητισμό. Δεν ε, ε, ασχολούμαι με το θέμα αυτό. Λυπάμαι, δεν μπορώ να σας δώσω μία απάντηση. Βεβαίως θα πρέπει να είμαστε άρτια προετοιμασμένοι και με το δικό σας input θα είμαστε ακόμα καλύτερα προετοιμασμένοι. Πρέπει να υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος με τους πολίτες και μέσω του αθλητισμού και βεβαίως ε, προσλαμβάνει ο αθλητισμός όλο ένα και ε, ευρωπαϊκότερη διάσταση με την αγορά παικτών και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια τα οποία έχουμε καταγράψει και θα επανέλθουμε όταν ε, υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε το σωστό άνθρωπο για τους πολίτες. Ε, είσαστε, έχετε μία πολύ ανοιχτή προσέγγιση. Θα λάβετε υπόψη αυτά που είπατε οι συνάδελφοι. Ε, υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Ε, ο εισηγητής έκανε ό,τι μπορούσε. Θα είμαστε λοιπόν σε επαφή Κυρίες, ε, κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώσαμε και τα διάφορα πριν ε, από αυτή τη συζήτηση, οπότε ολοκληρώσαμε την μερίστα διάταξή μας. Σας ευχαριστώ για τη συζήτησή μας. 5 Οκτωβρίου η επόμενη συνεδρίασή μας στις 3 το μεσημέρι. Δευτέρα είναι έτσι και μετά και την επακολουθή Τρίτη, 6 Οκτωβρίου στις 9 το πρωί. Ευχαριστώ και τους Ερμηνείς ε, και έχουμε τελειώσει από τώρα. Ωραία, γεια σας.